ανακοινώσεις. Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, σήμερα θα ψηφίσουμε σχετικά με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Για να επιτρέψουμε σε όλα τα μέλη να παραστούν με την κάρτα της ψηφοφορίας, οι ψηφοφορίες θα ξεκινήσουν στις 17 ακριβώς, στις 5 η ώρα. Ακριβώς. Εάν ε, συνεχίζεται κάποια συζήτηση εκείνη την ώρα, θα διακόψουμε την συνεδρίαση στις 16.55 προκειμένου να συνεχιστεί η συζήτηση μετά από το πέρας των ψηφοφοριών. Πριν από τις τέσσερις ψηφοφορίες επί της μεταρρύθμισης θα δώσω τους λόγους τους εισηγητές ε, για μια σύντομη τελική παρουσίαση. Σύντομη τελική παρουσίαση. Τονίζω, δεν θα υπάρξει συζήτηση. Υπενθυμίζω πως ακόμα και αν θα πρέπει τυπικά να ε, κάνουμε τέσσερις χωριστές ψηφοφορίες, η μεταρρύθμιση αποτελεί ένα συνολικό πακέτο. Ως εκ τούτου, εάν στην ε, ε, περίπτωση που απευχόμεθα ένας από τους τέσσερις φακέλους απορριφθεί, να γνωρίζετε ότι το σύνολο της μεταρρύθμισης θα τεθεί σε αμφισβήτηση. Σας υπενθυμίζω ότι η σημερινή μας συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω web stream και ότι η διερμηνία είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες ε, της Επιτροπής μας. Ωραία, περνάμε στο σημείο 4 της μισής διατάξεως, ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων ε, της Επιτροπής Γεωργίας το 2014. λάβετε υπόψη σας το, το χρονοδιάγραμμα το οποίο και δεχόμαστε. Βλέπω τη συνάδελφο Μαρία Γκάμπριελ που βρίσκεται ανάμεσά μας, περνάμε στο σημείο 5 της διατάξεως, τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου για το μέλη. Η συζήτηση επί της νομοδότησης ε, της κυρίας Γκάμπριελ για το ζήτημα που αφορά στο μέλη η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι ε, επί της αρμόδια. Το Συμβούλιο πρότεινε μια περιορισμένη τροποποίηση της οδηγίας του 2001 για να διευκρινίσει ε, τον όρο τους, ε, του, της γύρης ως φυσικού στοιχείου όπως είχε ε, λάβει υπόψη και το δικαστήριο στην υπόθεση Μπαμπλοκ, υπόθεση κάθε του 9. Αυτό, αυτό λοιπόν το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον των μελισσοκόμων. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια και υπενθυμίζω ότι η προθεσμία κατάσταση απολογιών έχει οριστεί η 7η Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Παρακαλώ Μαρία. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω υπενθυμίζοντα ότι η πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2110 του Συμβουλίου σχετικά με το μέλη είναι τεχνική φύση, αλλά η έγκρισή του, η απόρριψή του θα είχε κάποιες συνέπειε. Πρώτα απ' όλα γνωρίζουμε πως το ζήτημα να ξέρουμε αν η γύρις θεωρείται ως ένα ε, συστατικό φυσικό στοιχείο είναι ένα ζήτημα περίπλοκο και γι' αυτό το είδαμε μετά από επανειλημμένες ε, ε, δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης ε, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει και πολεμική. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να μακρηγορήσω κάπως προκειμένου να εξηγήσω στους συναδέλφους τι διάφορες ενημερώσει που έλαβα μετά από πολλές συναντήσεις που είχα με την Κομισιόν, τους μελισσοκαλλιεργητές, συμπεριλαμβανομένου και τον εισηγητή της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Σε ό,τι με αφορά να πω ότι καταρχήν εξέτασα αυτή την πρόταση από την προκειμένου να μην ε, ξεχαστούν οι επιπτώσεις που θα έχει στον τομέα το ενδιαφέρομενου κλάδου, δηλαδή της πελισσοκαλλιέργειας. Ε, ε, ο στόχος της Κομισιόν είναι να διευκρινίσει περαιτέρω την οδηγία 2110, οδηγία για το μέλι, αναφέροντας ότι το, γύρι είναι ένα συστατικό του μελιού και όχι ένα συνθετικό στοιχείο. Αυτό αποφασίστηκε το δικαστήριο στην απόφαση, στην υπόθεση Μπαμπλόκ. Αυτός ο ορισμός του 2013 213 ότι κάθε συστατικό θεωρείται ως, μάλλον τα συστατικά θεωρούνται όλα όσα χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία ενός ε, τροφίμου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της πρόεδρης της Κομισιόν που αντικαθιστά την προηγούμενη ε, διαδικασία της επιτροπολογίας της οδηγίας ε, με, για το μέλη μέσω της επιτροπολογίας το άρθρο, ε, το άρθρο 290 της, ε, συνθήκης. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων μεταξύ δικαστηρίου και κομισιών. Η αναφέρει ότι το ε, γύρι είναι ένα φυσικό συστατικό, ε, φυσικό, ε, φυσικό στοιχείο, διότι εισέρχεται στην, στο, στην κυρίθρα και ενώ το δικαστήριο τονίζει ότι όταν γίνεται φυγοκέντρηση κατά την διαλογή του μελιού, τότε υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθεί αυτό το, αυτή η γύριση και στους χώρους αποθήκευσης του μελιού. Γι' αυτό λοιπόν το γύριση η οποία περιέχεται στο μέλι αυξάνεται μέσω της διαδικασίας της φυγοκέντρησης. Γι' αυτό λοιπόν και συνέλεξα πολλές προφορίες χάρη σε συζητήσεις ε, επί του θέματος. Το πρώτο ζήτημα αφορά το πρώτο θέμα, ότι δηλαδή οι γύρις ε, είτε, ε, ότι είτε βρίσκεται, βρίσκεται, ότι βρίσκεται στο μέλι ε, εκ, εκ, εκφύσεως οι μελισσοκαλλιεργητές δεν προσθέτουν γύρι και άρα η πρόταση της Κομισιόν προσεγγίζει περισσότερο τα, την πραγματικότητα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θίγει η πρόταση αφορά την επισήμανση και τι τεστ δοκιμές. Πρώτον, ο ορισμός της γύρεως ως ε, συνθετικού θα έπρεπε, συστατικού συγγνώμη, θα έπρεπε να ε, γίνουν κάποιες δοκιμές αλλά να αναφέρεται και στην επισήμανση. Το, σύμφωνα τώρα με την Κομισιόν, το οι γύροι θα πρέπει σύμφωνα με την οδηγία 213 να μην θεωρηθεί ως συστατικό και να μην αναφέρεται στον κατάλογο των συστατικών. Γι' αυτό λοιπόν έτσι μάλλον καταλήγουμε στο κεντρικό θέμα που μας οδηγούσε στο θέμα της επισήμανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι έχουμε έναν κανονισμό ο οποίος αναφέρει πως όταν υπάρχει γενετικά τροπομενός οργανισμός στα προϊόντα θα πρέπει να είναι κατώτερο από 0,09%. Αυτό σημαίνει πως αν η πρόταση της Κομισιόν δεν γίνει δεχτή, τότε η ποσότητα της γύρεως γενικά τροποποιημένης ε, για να τηρήσει το όριο του 0,9% θα πρέπει να θεωρηθεί ως ε, ποσοστό συνολικής γύρης και όχι ένα ποσοστό της ε, συνολικής ποσότητας του μελιού. Εάν το όριο του 0,9% εφαρμόζεται στο, στο στη γύρι ως ε, συνθετικό υλικό, τότε θα θεωρηθεί ότι θεωρείται ότι θα πρέπει να αναφέρεται όχι στη συνολική ποσότητα του μελιού. Εξάλλου, αν η πρόταση της Κομισιόν γίνει δεχτή τότε είναι ελάχιστα δυνατόν το, η παρουσία της γύρεως ε, στο μέλι θα πρέπει δεν θα πρέπει να αναφέρεται στην ε, ετικέτα διότι θα βρίσκεται κάτω από το 0,9% για τη ε, νομοθεσία που αφορά τις γενικά τροποποιημένους οργανισμούς. <clears throat> Τώρα. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως ε, βρισκόμαστε πολύ μακριά από το όριο του 0,9%. Στα τέλη του Μαΐου 2013 δεν υπήρχε εξάλλου καμία, ένας τρόπος για εξέβραση των καταλλήλων ποσοστών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι απαιτήσει για την ε, ετικέτα. Εάν τώρα βασιστούμε στα τεστ, τότε θα πρέπει να κατασταθέσω ότι οποιαδήποτε και είναι η μορφή του τεστ που θα γίνεται και αν αυτό το τεστ καταστεί υποχρεωτικό, τότε θα δημιουργήσει υψηλέ επιβαρύνσεις για τους παραγωγούς και θα είναι ως εκ τούτου με λησοκόμοι αυτοί που θα, θα υποστούν τις επιπτώσεις. Θα έχουμε λοιπόν αρνητικό αντίκτυπο άμεσο στους ε, μελισσοκόμους έχουμε και έμεσες επιπτώσεις. Θα επιστρέψω την προσοχή σας στο γεγονός ότι γενικά το μέλι θεωρείται ως ένα φυσικό προϊόν και υγιές. Υγιεινό, Εάν το μέλι λοιπόν φέρει στην ετικέτα την σήμανση γενικά τροποποιημένου οργανισμού θα ε, επηρεάσει την ε, αγορά του μέλιου. Το όριο του 0,9% ισχύει για τα για τους βιολογικούς καλλιεργητές και είναι απαραίτητο να, βρεθεί, να ληφθεί υπόψη ότι αν λάβουμε υπόψη ότι η γύρι είναι συστατικό θα αποφύγουμε την άνηση μεταχείριση ανάμεσα στους παραγωγούς και τους ε, παραγωγούς βιολογικών προϊόντων. Αυτό δεν συμβαίνει αν ακολουθήσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Υπάρχουν και άλλες τρεις του θέματος που θα μπορούσαν να συζητηθούν. Υπάρχει το ζήτημα της ε, επιστήμικης ασφάλειας ε, σε ό,τι αφορά την επιστήμικη ασφάλεια η πρόταση της Κομισιόν δεν θα φέρει επιπτώσεις ε, επί της, για την ασφάλεια του μελιού διότι θα υπόκειται στους κανόνες για τα γενετικά του οργανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι εάν <clears throat> δεν είναι δυνατόν η εμπορία του είτε παράγεται στην Ευρώπη είτε σε τρίτη χώρα. Έτσι καταλήγουμε στο θέμα των τρίτων χωρών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε ότι κάποιοι μελισσοκόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι η εκτίμηση του δικαστηρίου σε σχέση με αυτήν τον καλλιεργητών τρίτων χωρών όπου ε, υπάρχουν γεννητικά τροποποιημένοι οργανισμοί, τότε θα υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση. πως το εξηγήσαμε, δεν υπάρχει καμία μέθοδος προκειμένου να ποσοτικοποιήσουμε το γενικά τροποποιημένο γύρι σε σχέση με την συνολική γύρι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να εφαρμόσουμε διατάξεις σχετικές με την σήμανση, ακόμα και αν ε, γύρι ήταν συστατικό. Επίσης, έχουμε εδώ και το θέμα της συνύπαρξης ε, Εάν κάποιοι συνάδελφοι επιθυμούν να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να επιμείνω το γεγονό ότι η συζήτηση για τροποποίηση τη οδηγία ε, περιμελιού δεν θα πρέπει να ε, δημιουργήσει σύγχυση με την συζήτηση για την συνύπαρξη. Δεν υπάρχει θέμα για συνύπαρξη σε κάθε χώρα. Έχουμε λοιπόν, γνωρίζουμε μάλλον ότι θα ήταν απαραίτητο να δημιουργήσουμε ζώνες αποκλεισμού της ε, διαδικασίας ε, φύτευσης οργανισμών γεννητικώς τροπημένων που θα πρέπει να ε, βρίσκονται σε απόσταση από 1 έως 10 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε και κανόνες που θα οριστούν και θα εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θα ήθελα να ε, στυλ, διότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το 12 2005 κράτη ε, καλλιεργούσαν σε εμπορική κλίμακα τις γενετικά τροπημένους κανονισμούς και είναι Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία και Σλοβακία. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια βεβαιότητα για την καλλιέργεια γενετικώς οργανισμών και μπορεί να συζητηθεί το θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά νομίζω πως εδώ θα είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε στην πρόταση όπως έχει σήμερα και μας επιτρέπει να ε, μιλήσουμε για, φυσικό συστατικό και όχι συνθετικό, ε, ως, συστατικό. Ε, συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα επί το οποίο δεν θα πρέπει να φυστούμε κόπον για να αποφύγουμε οποιαδήποτε χειραγώγηση του ζητήματος. Ευχαριστώ εκ των προδίων των συναδέλφων σου για τη συνεισφορά τους ή για τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ωραία, ευχαριστούμε Μαρία Γκάμπρια. Δώσουμε το λόγο στους τρεις εγγραμμένους. Άγνιου, πρώτος. I'm worried, Chairman, you use my Christian name for the very Πρώτη φορά με λες με το μικρό μου πρόεδρε. Ελπίζω να μην αρχίσουμε να γινόμαστε πολύ κολλητοί. Και να λοιπόν που περνάμε σε κάποιες από τις αποχρώσεις της αγγλικής γλώσσας, γιατί πριν από κάποια χρόνια συζητούσαμε αν θεωρούνταν τροφή ή ε, κατασκεύασμα, ή παρασκεύασμα μάλλον, το κέικ και το μπισκότο. Μέχρι που κάποια στιγμή κάποια επιτροπή το ξεδιάλεξε το ζήτημα. Και αποφάσισε ότι το ένα ήταν παρασκεύασμα και το άλλο μπισκότο. Και τώρα μας λέτε και το άλλο το τροφή. Και τώρα μας λέτε ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ Επιτροπής και Δικαστηρίου για το εάν είναι μέρος ή συστατικό του μελιού το, ή γύρι. Ενώ ε, ο ένας λοιπόν λέει το ένα και άλλο το άλλο και σας δίνεται ακόμη μια τρίτη απόχρωση, η, η λέει ότι είναι συστατικό του μελιού και πολύ θα χαρώ να δω να μεταφράζονται όλα αυτά σε τόσες πολλές γλώσσες. Το θέμα πάντως που τίθεται είναι τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς βρίσκεται μέσα στο μέλι. Γιατί δεν βρίσκεται μόνο μέλι, αλλά πάρα πολλά άλλα πράγματα, ε, όπως κυρίθρα, γύρι, ε, αυγά, ε, και πολλά άλλα πράγματα τα οποία προτιμώ να μην γνωρίζω και θα ήθελα να ελπίσω ότι θα είναι σε περιολάχιστες ποσότητες. Τώρα, αν επιδεινώσουμε την κατάσταση μιλώντας και για γενετικά τοποποιημένους οργανισμούς, ίσως είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα, γιατί και το φινικέλαιο είναι ε, γενετικά τροποποιημένο. Αυτό τουλάχιστον που χρησιμοποιείται στον Καναδά για την παρασκευή μελιού. Εμεί τέτοια πράγματα δεν έχουμε, αλλά μπορεί και να έχουμε, γιατί και στην Αγγλία υπάρχει ένα φινικέλιο που λέγεται υβριδικό και δεν φαίνεται να είναι προϊόν της μητέρας φύσης. Τροποποιημένο δεν είναι. Α, να τα που Δηλαδή, σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του, θα ο τέλος να λέμε «Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, δοκίμασέ το, όποιος βάλει το δάχτυλο μέσα στο μέλι, ξέρει». E Ευχαριστώ. Ρέμπερ και μετά Μάρτιν Όσλινγκ. Από την Άλτε καλωσορίζουμε την πρόσκληση της Ευρω... την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ την κυρία Γκαμπριέλ για την πολύ σαφή παρουσίαση. Η γύρι είναι φυσικό συστατικό και όχι επιπρόσθετη ουσία. Είναι ένα από τα λίγα φυσικά προϊόντα που δεν μπορεί να ανασυσταθεί, να κατασκευαστεί από τον άνθρωπο. Εάν ακολουθήσουμε τις προτάσεις για καταγραφή ως έκτακτης της παρουσίας της γύρης, μόνο να παραπλανήσουμε τον καταναλωτή μπορούμε και να τον αποτρέψουμε την κατανάλωση μελιού. Το δικαστήριο λόγω της φυγοκέντρης από ό,τι φαίνεται καταλήγει στην ασφαλμένη άποψη ότι μπορεί να υπάρξει μέλη και χωρίς γύρι. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό, διότι η γύρι βρίσκεται μέσα στο μέλι λόγω της φυσικής αυτής διαδικασίας ε, που έχει να κάνει με την ε, συλλογή από τη μέλισσα του μελιού των λουλουδιών. Άρα λοιπόν και στον ε, κόντεξ αλιμεντάριους και στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να πούμε ότι είναι καταγεγραμμένος φυσικό συστατικό του μελιού. Δεν μπορούμε να το συμπεριλάβουμε σε έκτακτα ή συμπληρωματικά συστατικά ή πρόσθετες ουσίες. Αυτό θα μας οδηγήσει σε πολλά προβλήματα και ενδεχομένω προσφυγές σε πέδο ΠΟΕ και στη δυσκολία στη σχέση μας με τρίτα κράτη. Η κυρία Γκαμπριέλ αναφέρθηκε στο ζήτημα του υπολογισμού της ε, παρουσίας γύρι σε περίπτωση γενετικά ομιλεί βέβαια για ελάχιστες, προϊόντων ή οργανισμών καλύτερα. Αυτό ομιλεί βέβαια για ελάχιστες, απειροελάχιστες ποσότητες. στην τελευταία ανάλυση η καταγραφή του μη γενετικά τροποποιημένου, η γύριση από μη οργανισμούς, ε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση και δεν μπορεί ο μελισσοκόμος να βεβαιώσει για την ύπαρξη ή ανυπαρξία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην γύρη, γύρη προερχόμενη από τέτοιου. Θα δυσκολεύσουν λοιπόν πολύ τα πράγματα εάν ζητήσουμε να καταγράφεται αυτό, να αναγράφεται αυτό στη συσκευασία και θα έχουμε σχολές προβλήματα και σε επίπεδο δικαστηρίου. Το μέλι λοιπόν που έχουμε στην Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό προέρχεται και από τρίτα κράτη, αλλά σε αυτή τη διαδικασία της αγωγής έχουμε πολύ μεγάλη παρουσία μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα αυτών των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την συσκευασία και ε, που ως εκ τούτου βρίσκονται θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη ε, θέση εάν επιδεινώσουμε την, την περιγραφή, υποβαθμίσουμε την περιγραφή του μελιού. Ε, από την άλλη πρέπει να προσέχουμε βέβαια να μην ε, επιτρέπεται η ανάμιξη με, την, ε, με ζάχαρη ή άλλες γλυκαντικές ουσίες του, του καθαρού μελιού γιατί πρέπει να προστατεύσουμε βέβαια το καθαρό μέλι και να αποφεύγουμε να παρασυρώμαστε σε συζητήσει για του τροποποιικά οργανωμένους οργανισμού, τροποποιημένου οργανισμού. τελευταία ανάλυση δεν έχει καν θέση εδώ. Ευχαριστώ, Χόισλινγκ. Και μετά η Επιτροπή. Δεν με ξαφνιάζει η μεγάλη αυτή οντάντ μεταξύ των δύο συναδέλφων που μίλησαν τελευταίοι. Που βέβαια ξεχνούν την ουσία της συζήτησης. Το ότι δηλαδή με την πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταφεύγει σε ένα τέχνασμα. Δεν μας βολεύει η συζήτηση για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και υπεκφεύγουμε με την δημιουργία ενός νέου νομικού πλαισίου που μας επιτρέπει να κλείσουμε ή να αποκλείσουμε καλύτερα τη συζήτηση για το δύσκολο θέμα του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Είναι μάλλον αστεία αυτή η πρόταση της Επιτροπής και έτσι πρέπει να την αξιολογήσουμε. Εν τέλει, θα είναι εις βάρος του μελισσοκόμου, ο οποίος βεβαίως, θα μπορεί, βεβαίως και μπορεί πρακτικά να εγγυηθεί ότι το μέλι του είναι καθαρό, όπως και η γύρι του, καθαρό από γενετικά τροπημένους οργανισμούς και αυτό θα σας εξηγήσω πώς γίνεται, είναι πάρα πολύ απλό με συγκεκριμένους κανόνες αποστάσεως είναι πολύ απλοί κανόνες αν θέλει κανείς να κάνει συζήτηση. Και χάρη σε αυτούς τους κανόνες μπορεί να εξασφαλιστεί αξιό, ε, ε, αξιόπιστη αναγραφή περί, μη περί απουσίας γενετικά τροπημένων οργανισμών. Αυτό είναι που άλλωστε χαιρετίζει στην πλειονότητα του, το, στην πλειονότητα των μελών του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτό μας λέει όταν σημειώνει ότι είναι ένα φυσικό προϊόν και δεν θα πρέπει να αναμεγνύεται ή να παρουσιάζει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Τώρα βλέπουμε να διαφεύγει η συζήτηση από αυτή την ουσία. Ε, φαίνεται να γίνεται αποδεκτή μια τυχαία επιμόρυνση, μια μικρή έκταση επιμόρυνση και εν τέλει φαίνεται ότι οι μελισσοκόμοι θα ε, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, εάν θέλουμε να είμαστε σαφείς, είναι δεδομένο ότι μπορούμε να έχουμε μέλη χωρίς γενετικά τρομμένους οργανισμούς. Υπάρχουν χώρες όπως η Αυστρία που έχει ήδη τέτοιου είδους ε, νομοθεσία και έχει ορίσει ότι η απόσταση, η ακτίνα μπορεί να διανύσει ε, μία μέλισσα πετώντας είναι τόση και ως εκ τούτου μέσα στην, ε, ε, σε μια τόση ακτίνα αποστάσεως από τις κεψέλες δεν μπορεί να υπάρχουν γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και ανάλογα γίνεται η αναγραφή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να λέμε ότι δεν είναι δυνατό αυτό. Έχετε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ασφαλώς και σε όγκο κυρίως, αλλά όπως έχει αυτή η έκθεση δεν μπορεί να γίνει δεκτή από εμάς. Ευχαριστώ όλους τους αδέλφους. Ο κύριος Έρικ Πότλετ, εκ μέρους της Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η ιστορία με τις γάματα φωμικρών είναι κάτι το οποίο συζητάτε συνεχώς στην Επιτροπή σας και σε άλλες επιτροπές στο Κοινοβούλιο και είναι ένα θέμα που εδώ και πολλά χρόνια συζητείται συνεχώς. Εμείς εδώ θέλουμε να τιμήσουμε την εισηγήτρια την κυρία Γκαμπριέλ και να πούμε ότι ίσως δεν είναι η στιγμή κατάλληλα να μιλήσουμε για την συνύπαρξη. Η Κομισιόν λοιπόν για να μην παίζουμε την κολοκυθιά αποφάσισε να να αποφασίσει για αυτό το θέμα και να πει ότι η γύρι δεν είναι ασυστατικό αλλά ένα φυσικό χαρακτηριστικό φυσικό στοιχείο του μελιού. Και όπως είπε η κυρία Καμπριέλ, ο μελισσοκόμος δεν προσθέτει γύρι θελημένα εκτός και βεβαίω αν θέλει να κάνει μια απάτη όπως γίνεται και με την κράμβη ας πούμε. Αλλά σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει αποτελεί απάτη και δεν νομίζω ότι αυτό το συζητάμε όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις. Θεωρούμε ότι το πνεύμα εδώ του Αρμπαμπλοκ τηρείται της Μπότσα Αρμπαμπλοκ τηρείται θέλουμε όμως να τονίσουμε ότι αν υπάρχει μέλη το οποίο είτε παρασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε προέρχεται από τρίτε χώρε το οποίο περιέχει γύρι, τροποποιημένη, μη εγκεκριμένη, τότε αυτό δεν μπορεί να διατεθεί στο εμπόριο. Στα σύνορα λοιπόν θα επιστραφεί στην χώρα προέλευσης. Αν περιλαμβάνει τώρα γύρι από μη εγκεκριμένο τροποποιημένο οργανισμό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα για τα υπόλοιπα, για την υπόλοιπη έκθεση, Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και χαιρετίζουμε την εργασία της κυρίας Γκαμπριέλ που εργάστηκε σε ένα τόσο δύσκολο τομέα. Τομέα που όπως είπε και η ίδια προκαλεί έτσι έντονες συζητήσεις και πάθη. Και ευθυγραμμισόμαστε και αποδεχόμαστε τη γραμμή της εκθεσής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στην συναδελφό μας την κυρία Καμπρίελ. και μετά πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους αδέλφους που σχολίασαν και συνέβαλα στη συζήτηση. Να ευχαριστήσω και την Κομισιόν που από την αρχή ήταν ανοιχτή για διάλογο. Είχαμε τακτικό και επικοδομητικό διάλογο, κάτι το οποίο επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε το θέμα χωρίς να υπάρχουν συναισθήματα που θα κυριορχούσαν στη λογική. Και αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους μελισσοκόμους. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που επέμειναν στο γεγονός ότι θα πρέπει να συγχαίουμε κάποιες συζητήσεις και κάποια θέματα συμπεριλαμβανομένων και στρέφοντας προς την κυρία Βρέσλινγκ. Ελπίζω να αλλάξουν κάποιες γνώμες μετά από την εις ανάγνωση της νομοδότησης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να εξετάσουμε την απήχηση που έχει αυτή η γνωμοδότηση και να μην δούμε μόνο την προτάση της Κομισιόν σε σχέση με το μέλη και να το προσεγγίσουμε ως κάτι που αφορά πολλές χώρες οι οποίες δεν έχουν εφαρμόσει ακόμα την οδηγία που περιλαμβάνει ένα πεδίο εφαρμογή για γεννητικά τροποποιημένου οργανισμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο τη τωρινή οδηγία. Πάντω όλα αυτά, ξαναλέω, είμαι ανοιχτή, είμαι δεκτική και ευχαριστώ όλου του συναδέλφου που συνέλαβαν στη συζήτηση με τροπολογίες και με τις απόψεις τους ώστε να δημιουργήσουμε να σχηματίσουμε μια σχέση του Κοινοβουλίου που δεν θα τροφοδοτείται μόνο από πολεμικές οι οποίες είναι χειραγώγησης αλλά θα μεριμνά για το συμφέρον και την προστασία των μελισσοκόμων που και αυτοί βεβαίως θα πρέπει να πράξουν τα δέντα προς την δική τους κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Κάπριλ. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο, στο έκτο τη ημέρα τη διάταξη. Βλέπω ότι ο κύριο Σιλβέστρη είναι εδώ, ανάμεσά μα. Πάμε λοιπόν στην παραγωγή και διάθεση, διάθεση φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά. Ένα λεπτό περιμένετε, μην κουνηθείτε. Ναι, ναι, δεν δε, δε, δε κουνιέμαι, Πρόεδρε. Πρόταση τη Κομισιόν, λοιπόν, σε σχέση με το φετικό αναπαραγωγικό υλικό. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η πρόταση αυτή τη οποία είναι εισηγητή ο κ. Σιλβέστερ, είναι τμήμα του νομοθετικού πακέτου για την υγεία των φυτών και των ζώων και που συζητήσαμε στην προηγούμενη μα συνεδρίαση. Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό αποτελεί έναν κύριο παράγοντα βασικό για τις επιχειρήσεις, για την υγεία, για τη γεωργία. Υπάρχουν πάνω από 7.000 επιχειρήσεις οι οποίε είναι σχεδόν όλες μικρομεσαίες που είναι ενεργές στον τομέα αυτό. Έχουμε πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη στον τομέα αυτό. Η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά αυτό το θετικό αναπαρικό υλικό και τη διάθεσή του βασίζεται κυρίως σε δύο πυλώνες. Την εγγραφή, την αναγραφή μάλλον των ποικιλιών και τις συγκεκριμένες οδηγίες που έχουν βγει σε σχέση με αυτό το φυτικό υλικό. Τώρα, το σχέδιο πρόταση του κ. νομίζω εδραιώνει αυτές τις προτάσεις και τις οδηγίες οδηγώντας εδώ 12 οδηγίες που υπάρχουν και που έχουν οδηγήσει σε κάποιο κατακαιρματισμό και σε διχογνωμία στι χώρε μέλη. Γι' αυτό ακριβώ υπάρχει ανάγκη εναρμόνιση. Και αυτό ακριβώ το λόγο, δίνω το λόγο αμέσω στον κύριο Σιλβέστρη και βεβαίω μετά έχουμε τη συζήτηση. Σέρτζο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για αυτή την εισαγωγή που νομίζω συνοψίζει τέλεια το πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται η συζήτηση για την έκθεση που αρχίζουμε να συζητάμε σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο συζητητής της πρότασης για το φυτικό αναπροϊκό υλικό θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις γενικές γραμμές αυτής της πρότασης. Το θέμα είναι περίπλοκο και αρκετά τεχνικό, όμως είναι κεφαλαιόδους σημασία, επειδή όπως υπενθύμισε ο Πρόεδρος αποτελεί την βάση ολόκληρης της ε, γεωργικής παραγωγής. Έχει λοιπόν μεγάλες ε, επιπτώσεις στην βιωσιμότητα και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. 7.000 επιχειρήσεις, 50.000 θέσεις εργασίας και κυρίως η ανάγκη απλούστευσης της ζωής και της δουλειά των επιχειρήσεων που δρούν στον τομέα αυτό και που σήμερα θα πρέπει να χαθούν στο δέδαλο 12 οδηγιών που τελικά θα συμπλέψουν, θα συγχωνευτούν σε μια νέα νομοθετική πράξη. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη απλουστευτική δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε που για κάποιες περιπτώσεις ανάγεται στα μέσα της δεκαετίας του 60. Παροχημένη και κατακαιρματισμένη λοιπόν νομοθεσία που όταν είχαμε νέες ενδείξεις και νέες ανάγκες που υπαγορεύονταν από την, από την αγορά και από την τεχνολογία προχωρούσε. Αλλά ενημερωνόταν με διάφορε διάφορες ε, οδηγίες και όχι με μία ενιαία όπως συζητάμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα σχόλιο για το στόχο του κανονισμού που είναι κάτι το οποίο συμμεριζόμαστε. Αυτό που έλεγα προηγουμένω δηλαδή, το να κάνουμε πιο ευέλικτη και πιο ταχεία την νομοθεσία στον τομέα αυτό και θεσπίζοντας κάποιες νέες προτάσεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των μικρών γεωργών και των βιολογικών καλλιεργειών. Κάποια σύντομα εισαγωγικά σχόλια να σας κάνω. Καταρχάς να διευκρινίσω ότι αυτός είναι ένας κανονισμός όπου επουδενή δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τους ε, γάματα φόμικρων. Και ούτε αυτούς βεβαίως που είναι μικροκαλλιεργητές στα σπίτια τους ή σε μικρά χωράφια ή στους κήπους τους. Δηλαδή ο καλισμός αυτός δεν καλύπτει υλικό το οποίο προορίζεται σε τράπεζες γάματα φόμικρων και δεν αφορά βεβαίως τους μη επαγγελματίες, του ερδεχνές δηλαδή του τομέα αυτού. Όποιος λοιπόν δεν είναι φορέας επαγγελματικός στον τομέα αυτό δεν εμπλέκεται και δεν είναι αντικείμενο των διατάξεων του κανονισμού. Το κείμενο που συζητάμε λοιπόν σήμερα ακολουθεί μια ανάλυση εμπειρογνωμόνων και μελέτες και σχόλια που μπόρεσαν να υποβάλουν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι στον τομέα, διάφοροι μετά από έρευνες στη, της Επιτροπής από το 2007 και 2008 μέχρι το 2010. Αυτό που ανακύπτει μετά από διάφορες ε, συζητήσεις και επαφές που είχα με τους εκπροσώπους του κλάδου ότι η ισχύουσα δομή όσον αφορά αυτό το υλικό φαίνεται να ικανοποιεί τους πάντες. Δηλαδή έχουμε μία δομή με δύο πυλώνες που προβλέπει αφενός την αναγραφή της ποικιλία στον αναπαραγωγικού υλικού αφενός και αφετέρου την ένδειξη για μεμονωμένες παρτίδες που διατηρείται σε αυτό το κανονισμό. Δύο λόγια για την πιστοποίηση. Το ΒΑΟ η αναγραφή δηλαδή της επιχείρησης όταν έχει τα εργαλεία στη διάθεσή της για το υλικό πριν από τη διάθεσή του στην αγορά. Δεν θα πρέπει πια να περνούν από την ισχύουσα διαδικασία, αλλά απροστεύονται διαδικασίες και η έλεγχη από την αρμόδια αρχή. Νομίζω ότι αυτό που δεικνύει ότι η εν λόγω νομοθεσία έχει ως στόχο την πραγματική απλούστευση χρόνων και διαδικασιών. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο μία επαγορευμένη ανάγκη από την ύπαρξη ενός ενιαίου κειμένου, αλλά και από την ανάγκη ύπαρξης απλουστευμένων διαδικασιών. Επίσης και για την πιστοποίηση και για τους δασμούς μετά θα επιφυλαχτώ να καταθέσω κάποιες τροπολογίες για το κείμενο. Πάντοτε για το θέμα του ΒΑΟ, ΒΑΟ η αγρονομική αξία χρήσης θα πρέπει να είναι ικανοποιητική και βιώσιμη. Αυτό το τελευταίο κριτήριο αντιπροσωπεύει νομίζω μία καινοτομία σε σχέση με τα ισχύοντα. Και τα τελευταία άρθρα που το αφορούν, ιδιαίτερα αναφέρομαι στο 58 και 59 άρθρο του κειμένου, θα είναι καλό να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο κάποιων αλλαγών που θα σας προτείνω στη συνέχεια. Επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη επισκόπηση των κοινοτομίων που παρουσιάζει αυτός ο κανονισμός. Ιδιαίτερα όσον αφορά το 14 και το 36 άρθρο. Είναι οι δύο πυλώνες της ε, πρότασης που δεν περιλαμβανόταν στην ε, οδηγίες που καταγουνται με αυτό το νέο κείμενο, αποτούσαν όμως ε, αποκλήσεις και μάλλον παρεκκλήσεις που είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε το θέμα των μικρών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων οι οποίε μάχονται για την βιοπικιλότητα και παραγωγού και γιορού οι οποίοι πουλούν μικρέ ποσότητε. Μετά από πολλέ επαφέ με τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσα να σα πω ότι αυτά τα δύο άρθρα είναι τα άρθρα στα οποία συγκεντρώνεται, στα οποία επικεντρώνεται μάλλον το μεγαλύτερο μέρο των ανησυχιών και επί των οποίων αναπόφευκτα θα εστιάσει και η προσοχή της Επιτροπής μας μέσω κατάθεσης τροπολογιών. Η εντύπωση μου ότι η Κομισιόν έχει μείνει λίγο αόριστη όσον αφορά του καθορισμό των λεπτομεριών. Έχουμε ένα νέο τμήμα βεβαίω ε, νομοθεσία το οποίο είναι χαρτογράφητο, αλλά αφήσαμε στι κατεξουδότητε οι πράξει πάρα πολλά θέματα, ενώ αντίθετα όλα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην βασική πράξη. Τώρα για τις παλαιότερες ποικιλίε, οι οποίες ήταν τμήμα ήδη της ισχύουσας νομοθεσίας, το θέμα είναι εξίσου επίμαχο. Δηλαδή, θέλουμε να προβλέψουμε ελάφρυνση του διοικητικού γραφειοκρατικού φόρτου, όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα εφαρμοστικά. Τη στιγμή ιδιαίτερα που ζητάμε το υλικό, παρόλο που δεν θα πρέπει να υποβάλλεται στον τόση στο ΒΑΟ, θα πρέπει ούτως ή άλλως να αναγράφει στην σήμανση τον τόπο προέλευσης και παρόλο που, μάλλον είναι δυνατόν να διατεθεί παντού στο εμπόριο, σε οποιοδήποτε μέρος. Παρόλο που είμαστε υπέρ λοιπόν των σημάνσεων ε, ονομασίας προέλευσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε διακρίσεις για τους παραγωγούς για τους οποίους επανειλημμένως έχουμε θελήσει να προστατεύσουμε σε άλλε εκθέσει μα, αλλά για τα γάματα φόμικρον βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο. Δηλαδή, έχουμε ένα μικρό κομμάτι τη αγορά σήμερα που παρουσιάζουν όμω θέμα προέλευση, αλλά για ιστορικού λόγου δεν καλλιεργούνται πια. Και αυτό βεβαίω συνεχίζει να αποτελεί τμήμα μια μικρή ακόμα αγορά, αλλά ο γεωγραφικό περιορισμός προέλευση είναι δύσκολο να καθοριστεί. Όσον αφορά τώρα το import-export του αναπαραγωγικού υλικού στο 6 του κειμένου χαίρομαι για την βούληση της Κομισιόν να προβλέψει μια αναλογία του υλικού που θα εισαχθεί από τρίτες χώρες όσον αφορά την ποιότητα και την τήρηση των κανόνων. Επιτέλους, επιτέλους θα προσταταγώ. Όσον αφορά το θέμα των εξαγωγών, επιτρέψτε μου να κάνω να πω το εξή ότι θα πρέπει δηλαδή να βρεθεί μια περαιτέρω λύση ώστε για τους εξαγωγούς των σπόρων να μην υπάρχει πρόβλημα γραφειοκρατίας και κόστους. Και να επιθυμίσω από την ευκαιρία ότι από την ΕΕ ξεκινάει το 60% φυτών και σπόρων παγκοσμίω τομέας ηγέτης στην γεωργία μας, χάρη και στις προσπάθειες των επιχειρήσεων για βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Τέλος, για να φτάσω στο τέταρτο τμήμα και φτάνω μάλλον στο τέταρτο τμήμα του κειμένου από το 105 άρθρο και μετά όποτε αναλύουμε το δασικό αναπαραγωγικό υλικό δεν θα πω πολλά η ισχύουσα νομοθεσία νομίζω ότι εδώ έχει περιληφθεί καρμπών στον νέο κανονισμό μετά από έτοιμα βεβαίως και των εμπλεκομένων των προσώπων του, του κλάδου που εξέφρασαν και την ικανοποίησή τους όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία. Οπότε δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το τμήμα θα πρέπει να αλλάχθει, να τροποποιηθεί ουσιοδός στο κείμενό του. Τελευταίο σημείο, κάτι το οποίο αφορά την διαδρομή και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει η δουλειά μας. Η Επιτροπή ΕΜΒΗ ζήτησε και έλαβε την ε, κοινή αρμοδιότητα για επισημία σημεία αυτού του κανονισμού. Ιδιαίτερα η περιγραφή του επισήμου αναγνωρισμένου, παρεκκλήσεις από την στάνταρ τα, τα είδη τα οποία είναι προστατευμένα, οι ποικιλίε και αναγραφή τους, οι παρεκκλήσεις μικροεπιχειρήσεις και οι γενετικές, γενετικές βάσεις και τράπεζες. Αυτά. Τώρα βέβαια συνάδελφοι εγώ θα ακούσω με μεγάλη προσοχή προτάσεις και συστάσεις που θα ανακύψουν. Επειδή η δουλειά αυτή θα πρέπει να είναι κοινή και να καταλήξει σε μια κοινή αποδοχή. Για δύο λόγους. Πρώτος, το είπα στην αρχή της ομιλίας μου, επειδή το θέμα είναι πολύ σημαντικό και αποτελεί το σημείο κίνησης της Γεωργίας δηλαδή η διάθεση στο εμπόριο του φυτικού υλικού αποτελεί τη βάση του γεωργικού εμπορίου. Το υγιές φυτικό υλικό τη στιγμή που μάλιστα και η Ευρωπαϊκή Ένωση με ορίζοντα το 2020 μας ζητά να δουλέψουμε για την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα. Η διάθεση λοιπόν, η διαθεσιμότητα υλικού, φυτικού υγιούς είναι απαραίτητη ώστε να αποφευθούν πράξεις οι οποίες είναι κατά της ε, βιωσιμότητας και που πλήττουν την ίδια τη Ο άλλος λόγος για να προωθήσουμε την δουλειά μας είναι το ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε συμβιβασμούς και συνθέσεις γρήγορα, τότε θα τελειώσει η θητεία χωρίς να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει. Και αυτό βεβαίως θα οδηγούσε σε αποτυχία όσον αφορά την έγκριση, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση, τη έκθεσης αυτή. Γι' αυτό ακριβώ λοιπόν θα είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός στις παρατηρήσεις σας όλων και ελπίζω να ανακύψουν από εκεί στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν το ταχύτερο δυνατόν να κάνουμε την καλύτερη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ Σέρτζο. Τώρα προχωράμε. Διάφοροι συνάδελφοι μου στήσει το λόγο. Αν κατορθώσουμε να παραμείνουμε στο χρονικό όριο που έχουμε στη διάθεσή μα, θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε το σημείο προτού να περάσουμε στι ψηφοφορίε σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ΚΑΠ. Herbert Ντόρφμαν και Μάρτιν Όσλι. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο Σέρτζο Είναι ένα θέμα το οποίο επικρίθηκε πριν καλά-καλά βγει από την Κομισιόν. Ξέρουμε ότι ο Σέρτζο τόνισε το ζήτημα των σπόρων και των φυτών ε, παλαιών, εμπιστοσύνη που έχουν διαδοθεί μόνο τοπικά και αυτό προκάλεσε μια συζήτηση σοβαρή είμαι πεπισμένος πως ε, χρειάζεται να εξευρεθεί λύση. Όποιος χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιεί ή θέλει να φυτέψει ένα φυτό μιας τοπικής ποικιλία ή να χρησιμοποιήσει ένα σπόρο τοπικό θα μπορεί σίγουρα και θα πρέπει να μπορεί να το πράξει. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζει τον κίνδυνο που διατρέχει. Ο κίνδυνος είναι ότι το φυτό μπορεί να μην είναι υγιές και όλοι όσοι ασχολούνται με το ζήτημα αυτό τα γνωρίζει αυτά τα προβλήματα. Είναι περιττό να θέσουμε νέους κανόνες και περιττούς θα έλεγα, αλλά για το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής νέων φυτών και σπόρων το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία και η πιστοποίηση θα πρέπει να γίνεται κατανοητή ως κάτι που χρησιμεύει στους μεγάλους της αγοράς. Δεν θα πω παραπάνω διότι τους γνωρίζουμε όλοι. Εγώ προέρχομαι μια περιοχή που παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους φρούτων και όποιος αγοράζει από εκεί φρούτο θα πρέπει να γνωρίζει ότι αγοράζει την χη τον ψη ότι το φυτό είναι υγιές, εξάλλου όσοι παράγουν αυτές τις, ε, αυτά τα φυτά θα πρέπει σε περίπτωση λάθους να είναι υπεύθυνο. Αν αγοράζω ένα φυτό ή μια, ένα σπόρο για δίποτε ποικιλία και αν κάποιος μου το πουλήσει, μου δώσει κάτι το διαφορετικό, τότε θα πρέπει να είναι υπεύθυνο. Άρα υπάρχει και η υπευθυνότητα του παραγωγού σπόρων και φυτών. Η πιστοποίηση λοιπόν είναι τμήμα της ασφάλειας και δεν πρέπει να ξεχνάμε την επένδυση που κάνει ένας γεωργός για νέο φυτό. Εάν κάποιος φυτέψει ένα αμπέλι και μετά από πέντε χρόνια ανακαλύψει ότι δεν ήταν το φυτό που είχε αγοράσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές, αυτό που είχε ζητήσει, τότε έχει επενδύσει χρόνια εργασίας, έχει επενδύσει στον αγρό τον οποίο δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει για άλλους λόγους, είναι αυτό δεν είναι σπάνιο, συμβαίνει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και η πιστοποίηση για όλα τα φυτά, όλους τους σπόρους θα πρέπει να διέπεται από αυστηρούς κανόνες Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Χέρμπερτ, ο Μάρτιν Όσλιν και μετά η συνάδελφος Κάντεμακ. Μάρτιν. Γεια, μανεστε äh, Damen Ξέρετε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, μπορεί να κρύβονται καλές προθέσεις πίσω από την ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, αλλά έχουμε πολλές φορές αντιμετωπίσει το πρόβλημα να χάνονται αναπαραγωγικό υλικό μικρότερου μεγέθους και αγορές, ενώ επικρατούν μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως ε, προερχόμενες από το κλάδο της χημικής βιομηχανίας, και που επιβάλλουν αυτό που θέλουν ενώ εμείς προσπαθώντας να διαφυλάξουμε την ποικιλομορφία αγωνιζόμαστε και για την διαφύλαξη του αναπαραγωγικού υλικού. Έτσι λοιπόν Επιτρέψτε μου να διατυπώσω την εξής ένσταση. Όταν έχουμε μία μικρή μεσαία επιχείρηση, τα όρια που θα θεθούν ε, για την ε, διαφύλαξη του παραγωγικού υλικού δεν έχουν καμία αξία. Και αν θέλουμε να κάνουμε μια αν θέλουμε να εισαχάγουμε υψηλό επίπεδο προστασία, πρέπει και τα όρια να είναι υψηλά και αντίστοιχα να ξέρουμε τι επιδιώκουμε, γιατί με την απελευθέρωση του συστήματος, στην καταχώρηση ή την αδειοδότηση αναλόγως, μόνο μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές των μικρότερων επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και απαλλαγή τους από, το γραφειο, από τη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Εγώ νομίζω ότι κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Ωστόσο, ότι είναι τόσο υψηλές οι απαιτήσει για τις μικρότερες επιχειρήσεις δυσβάσταχτες, δυσβάσταχτες όπως τις ορίζουμε, που δεν δίνουν την ευκαιρία της επιβίωσης για επιχειρήσεις οι οποίες παραδείγματι δεν έχουν ε, προσανατολισμό προς τις εξαγωγές κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να επισημάνουμε ως κίνδυνο. Και αν ε, θέλουμε να συζητήσουμε και περισσότερο, να δούμε τι λέει, τι έλεγε μάλλον σε μια πρώτη της πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλει να υποστηρίξει τις εξαγωγές, τις οποίες βέβαια δεν θα δούμε να τις ε, αναπτύσσουν οι μικρότερες επιχειρήσεις. Αυτές οι 7.000 επιχειρήσεις λοιπόν για ποια αγορά παράγουν, για την ευρωπαϊκή κυρίως. Γι' αυτό και δεν πρέπει να τις ταλαιπωρούμε με περί τη γραφειοκρατία. Αυτή λοιπόν ε, η απέτηση για βιολογικά ανα, για βιολογικό αναπαραγωγικό υλικό, για καλή ποιότητα αναπαραγωγικό υλικό, νομίζω ότι είναι αυτή που θα πρέπει να προβληθεί από τον εισηγητή και όχι οι απαιτήσει και προσδοκίε τη μεγάλη βιομηχανία των φυτικών αναπαραγωγικών πόρων. Εάν ακολουθήσουμε την πρόταση επιτροπή, θα χάσουμε πολλέ από τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Και αυτό είναι ακριβώ που θα πρέπει να αποφύγουμε γιατί χρειαζόμαστε όχι τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ε, οι οποίες μόνο για λόγους μουσιακούς μπορούν να διαφυλάσσουν κάποιο αναπαραγωγικό ε, υλικό, αλλά εκείνες οι οποίες ζουν και εργάζονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, διατηρούν τη ζωτικότητά της και ταυτόχρονα αναπαράγουν το υλικό αυτό το φυτικό για λόγους παραγωγής και όχι για λόγους μουσιακούς. Ευχαριστώ κυρία Κάρνμπαχ. Ευχαριστώ και καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστώ τον ε, Πρόεδρο και τον συναλφό Σιλβέστρες για την ε, πρόσκληση και την ενημέρωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόταση για τον κανονισμό για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό όπως ονομάζεται έχει κάνει μια, ένα βήμα παραπάνω ε, και γνωρίζω από τους Γερμανούς συναδέλφους και τους Αυστριακούς ότι ακόμα και πριν να δημοσιευθεί επί η πρόταση αυτή είχε προξενήσει πολλές ανησυχίες και στις δύο χώρες και πολλές συζητήσει. Παρακαλώ λοιπόν την Επιτροπή να λάβει υπόψη και πολύ σοβαρά τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί. Να μην τις παραμελήσει. κύριος Χάισλινγκ έχει ήδη άλλωστε εξηγήσει σε λεπτομέρειες τα ζητήματα και καλό θα ήταν να μην υποχωρούμε πάντοτε σε αυτούς οι οποίοι έχουν το μεγάλο όγκο της παραγωγής στην, και, τον έλεγχο της, και να επιτρέπουμε να λάβουν και τον έλεγχο της βιοπικιλότητας. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει το υλικό αυτό το αναπαραγωγικό για τον καταναλωτή, για τη γεωργία, για την ανεξαρτησία του γεωργού από τις εταιρείες ε, διαχείρισης αυτού του υλικού. Αυτό θα, θα έπρεπε να είναι μάλλον το δυναμικό της πρότασης. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα άρθρα δεν εξυπηρετείται αυτός ο στόχος ικανοποιητικά. Πραγματικές βελτιώσεις του status quo είναι μόνο περιορισμένες και βλέπω ότι δυστυχώς ε, του ναντίον έρχεται νέα γραφειοκρατική επιβάλληση με την πρόταση αυτή. Υπάρχουν ειδικές οδηγίες οι οποίες ήδη καλύπτουν και συνθήκες διαφύλαξης και ε, τα είδη, οι οποίες είναι πιο ειδικέ και θα συνεχίσουν ασφαλώς να εφαρμόζονται. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να προχωρήσει αυτή η πρόταση και εμένα πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει να δούμε ο κλάδος παραγωγικός ε, στις διάφορους τομείς τι συνέπειες μπορεί να αντιμετωπίσει λόγω αυτής της ε, πρότασης. Καταρχάς η διαφύλαξη του αναπαραγωγικού υλικού παραμένει ένα σημαντικό, ένα σημαντικό κομμάτι αγοράς, μια νέα αγορά, νήσο όπως την ονομάζουμε και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διατυπώνει προτάσεις οι οποίες δεν θα βρουν συμφωνή την ε, διεθνή την κοινή γνώμη και βέβαια τους δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους της. Διερωτώμεθα τι είδους στόχους εξυπηρετεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γιατί δεν εξαιρούνται απολύτω οι ιδιώτες από το πεδίο εφαρμογή αυτού του κανονισμού, γιατί δεν γίνεται διερεύνηση σε δεχόμενες ιδιωτικές δραστηριότητες. Και θα ήθελα να αφαιρθώ στα εξή σημεία, ότι θα πρέπει να διαφυλάσει την ελευθερία για την επιλογή των φυτών και σιτηρών από τον καταναλωτή, αν δηλαδή θέλει να είναι παραδοσιακής παραγωγής ε, ή διαφορετικά τα προϊόντα που θα καταναλώσει. Ε, αν θέλει να είναι συμβατική σπόροι ή ε, ειδική και σπάνη. Και τώρα έχουμε τρεις και δεν νομίζω ότι εξυπηρετείται αυτός ο στόχος ικανοποιητικά. Τώρα έχουμε τρεις μεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο των, του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού των σπόρων που διαχειρίζονται το 50% της αγοράς και από αυτές περνάει τεράστιο ποσοστό των τροφίμων μας. Άρα και τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια της ε, προμήθειας τροφίμων, του φοδιασμού σε τρόφιμο, που θα πρέπει να είναι πρώτο μας μέλημα. Όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ιστορικό, αλλά και σε σχέση με τα αναπτυσσόμενα κράτη, θα πρέπει να το δούμε αυτό άλλωστε. Και ιδιαίτερα θα ήθελα όσο οι δημοκράτες να διεκδικήσουν μια καλύτερη προστασία του αναπαραγωγικού υλικού, του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, Ιδιαίτερα θα πρέπει να αφερθούμε στην προστασία των γενετικών πόρων και να ενισχυθούν οι κοινοφελείς πρωτοβουλίες των πολιτών κυρίως για το περιβάλλον, για τη βιοπικιλότητα και ως εκ τούτου θα καταθέσουν μια σειρά από τροπολογίες στους άλλους Και θα ήθελα να απευθύνω μια γενική έκκληση. Μίλης μου ότι έρχονται ευρωεκλογές μόνο ότι ο πολίτης και πολύ σωστά απαιτεί να αντιμετωπίζεται ο ίδιος και οι προσδοκίες του, οι ανάγκες του με σοβαρότητα. Αυτή η συζήτηση που ξέσπασε, ο δημόσιο διάλογο που ξέσπασε μόνο με την ανακοίνωση ότι θα κατευθεί πρόταση, ήδη δείχνει πόσο μεγάλη σημασία αποδίδει ο κόσμο και δείχνει επίση ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκλείσουμε την ανάπτυξη επιπλέον γραφειοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Άγνιου έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το θέμα αυτό για το αναπαραγωγικό υλικό δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη αναταρχή στον Ηνωμένο Βασίλειο, μάλιστα και στις, ε, ε, στην ώρα ερωτήσεων προς τον Υπουργό έγινε μεγάλη συζήτηση στη Βουλή αλλά και γενικότερα στην κοινή γνώμη. Έτσι λοιπόν στις γενικές διατάξεις υπάρχει πρόθεση για μια διάταξη η οποία θα λέει ότι η ιδιωτική ανταλλαγή σε είδος φυτικού αναπαραγωγικού υλικού αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Δεν πρέπει να διαγραφεί αυτή η πρόταση από την Επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλη τροπολογία μπορεί να κατατεθεί. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια για τους κυπουρούς της Βρετανίας, αλλά ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σαν στόχο να, συστάλει ακόμη, να, συστήλει ακόμη περισσότερο, περισσότερο την ε, λειτουργία και το πεδίο αυτή τη ε, διατάξεω. Ε, Όπω είπα, όμω ανησυχούν πάρα πολύ οι κυπουροί τη Βρετανία και αυτό παρακαλώ την Επιτροπή να με καθησυχάσει ω προ την υπόθεση αυτή. Εδώ έχουμε να κάνουμε την ανάκληση και αντικατάσταση από, ένα, από μια υπεροδηγία των 12 ήδη υπαρχουσών μας λέτε ότι, αυτός, ότι ο στόχος είναι της απλουστεύσεως, μα ασφαλώς και με την ε, ΚΑΠ έτσι είχατε ξεκινήσει και μιλούσατε για απλούστευση πριν από μερικά χρόνια, τώρα όμως ξέρουμε πολύ καλά που έχουμε φτάσει. Ε, you keep, Κύριε Ρόντουστ, ε, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει αναπτύξει αρκετές επαφές και συνομιλίες ο εισηγητής έχει συστήσει εντατικά με όλους τους εμπλεκομένους, ωστόσο παραμένουν κάποια ερωτηματικά. Και παρακαλώ τον εισηγητή γραπτός να δώσει απάντηση στις ερωτήσεις μου μέσα από την έκθεσή του. Πρώτον, μόνο για την εμπορική χρήση και αποκλειστικά στην χρήση μεγάλης κλίμακας, εμπορικής κλίμακας ε, θα περιοριστεί αυτό ε, το πεδίο εφαρμογή, ε, γιατί έχουν γραφτεί αρκετά συγκρουόμενα στοιχεία και δεν βλέπω πουθενά να υπάρχει αποσαφήνιση μέσα από το κείμενο. Δεύτερον, η ανταλλαγή φυτικού ή αναπαραγωγικού υλικού για ιδιώτες, μεταξύ ιδιωτών και πουρών και το καθεξής. Λέγεται ή ακούγεται εν γέννη ότι πρόκειται να παραμείνει ελεύθερη, αλλά πώς θα οριστεί αυτό, πώς θα γίνει στην πράξη και μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην πράξη πώς θα ισχύσει. Είναι καλό να γνωρίζουμε τι θα συμβεί και να συγκυρίζει και ο καθένας τι ισχύει. Και επίσης για τις ε, παραδοσιακά καλλιεργούμενες ποικιλίε θα παραμείνει ελεύθερη η αγορά ή θα υπάρχει δυνατότητα για την διεκδίκηση ε, δικαιωμάτων πραγματικής διοκτησίας ενδεχομένω και διπλώσματος εύρε τεχνίας. Αυτό φαίνεται ότι προς τα είναι τελικά. Επίσης, υπάρχει η ανάγκη να δοθεί ένας σαφής προσδορισμός για τις οικολογικές καλλιέργειες. Αυτό το έχει παραλείψει η πρόταση. Και μια τελευταία ερώτηση σχετική με τη διαφάνεια. Πώς θα οργανωθεί στο μέλλον ε, το ζήτημα της διαφάνειας ως προς τα δικαιώματα πνευματική διοκτησίας, ε, ενδεχόμενα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τις υβριδικές ποικιλίε, ε, λοιπές μεθόδους παραγωγής, καλλιέργειας πώς θα μπορεί ο κάθε ένας που θέλει να γίνει γεωργός ή καλλιεργητής ή απλός κυπουρός να χρησιμοποιεί αυτό το υλικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ρέιμερς, μετά ο κύριο Κόπουλο. Ευχαριστώ. Για την ερώτηση του κύριου Άκνιου. Είναι απλούστευση το να το να ρίχνουμε τα πάντα μέσα σε ένα κόρβανα και να, και να τα ανακατεύουμε όλα τελικά δεν γίνεται πολύ πιο περίπλοκο το σύστημα. Δεύτερον, βλέπω πάρα πολύ μεγάλο αριθμό κατεξουσιοδότηση πράξεων, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι σε άλλα νομοθετήματα. Και ως εκ τούτου ανησυχώ αγαπητοί Κομισιόν, μπορεί να είστε εσείς ε, ένας ε, υπερμεγέθης οργανισμός διαχείρισης, αλλά την νομοθεσία τον κάνει, την κάνει το Κοινοβούλιο και οι βουλευτές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει εμείς να αποφασίζουμε και να κρίνουμε πού είναι η ανάγκη κάθε φορά είτε να αναλάβει η διοίκηση κάποια ε, διαδικασία να την ολοκληρώσει, κάποια διατύπωση ή να γίνει η παρέμβαση νομοθετική. Αλλά εμείς πρέπει να το κρίνουμε αυτό. Επίσης από, όλο, από την όλη αυτή δέσμη μέτρων βλέπουμε να μην υπάρχει επαρκή κάλυψη σε περίπτωση ε, ζυζανίων και καραντίνα σε περίπτωση ζημιωγών οργανισμών. Ε, ο καλλιεργητής, γεωργός, ο οποίος πρώτος θα το εντοπίσει αυτό ε, το ζυζάνιο, κινδυνεύουμε να δούμε να μην το δηλώνει, να μην το καταγράφει, να μην το καταγγέλει, διότι κινδυνεύει ο ίδιος να υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά. αυτόν ο πρώτος στην αλυσίδα. Ε, εδώ λοιπόν θα πρέπει το σύστημα της καραντίνας να αναθεωρηθεί, ίσως και γενικότερα το σύστημα. Βλέπω ότι θέλει η Επιτροπή ένα πιο σύγχρονο σύστημα με ολογράμματα, με γραμμές, με συστήματα που θα επιτρέπουν μια πρόσκοπτη λειτουργία του ε, συστήματος καταγραφής και ίσως λιγότερα ε, έντυπα, αλλά πολλές φορές ε, μας δίνονται οι πληροφορίες μέσα σε ένα εγχειρίδιο το οποίο είναι αρκετά ογκώδες και άρα δεν έχει το στόχο της μείωσης κατανάλωσης χάρτου. Για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό με επιλεκτική ε, παραγωγή θα πρέπει να μην συμπεριληφθεί σε αυτόν τον ε, κανονισμό είναι ένα διαφορετικό σύστημα ανάπτυξης ε, ποικιλιών και ως εκ τούτου και δεδομένου ότι έχει και πολλά χαρακτηριστικά που εξαρτώνται από την κάθε περιφέρεια και το μικροκλίμα ή τις ιδιαιτερότητες της, δεν μπορεί να ε, γενικεύεται και να περνάει σε αυτόν τον κανονισμό. Εάν ας πούμε, σκεφτούμε ένα συγκεκριμένο είδος ελάτης που μπορεί να υπάρχει στη Βόρεια Γερμανία, αυτό δεν μπορεί να μεταφερθεί ε, με τη μορφή σπόρων και να φυτευτεί και να ευδοκιμήσει στην Αυστρία Φερρυπίν, γιατί τελείως διαφορετικές οι φυσικές συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ. Λουίς Κάπουλα Σάντος και μετά ο κύριος Ταραμπέλα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σιλβέστρης για την παρουσίαση που μας έκανε. Γνωρίζουμε ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και πολύ ευαίσθητο. Όλοι λάβαμε χιλιάδες ε, email γιατί είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε την κατάλληλη απάντηση. Όλοι γνωρίζουμε την ανάγκη ύπαρξης ενός μητρώου πιστοποίησης κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού μας βίου. Όλοι Είχαμε σχέση με φυτά τα οποία αγοράσαμε, ε, ήταν ασθενή και πολλές φορές ο αγοραστής δεν αγοράζει αυτό το οποίο επιθυμεί. Πολλές φορές ε, αγοράζει κάτι το διαφορετικό. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε τις απαραίτητες εγγύησεις ε, υγιεινής και ασφάλειας για τους γεωργούς και όχι μόνο, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε και την ε, γραφειοκρατία, ειδικά για τους ε, μικρούς ε, παραγωγούς, μικρούς καλλιτηγητές. Εγώ είμαι και ο εκ μέρους της ομάδας μου. Είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με τον εισηγητή σας για να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις και να συμβάσουμε τους λόγους αυτούς που προανέφερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι θέμα εμβληματικής σημασίας, ε, δημιουργεί συζητήσεις, αντιδράσεις, ίσως και υπερβολικές κάποιες φορές, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω από το στόμα της Κομισιόν που έκανε την πρόταση, εάν ε, οι όροι που χρησιμοποιούνται, δηλαδή διάθεση στην αγορά, αναφέρομαι στα αυτοτρια 3 της πρότασης, που περιέχει τους όρους θέση στην αγορά, διαθεσιμότητα στην αγορά, ότι αυτό σημαίνει την κατοχή εν ώψη της πώληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, δηλαδή της ε, ε, αγοράς εν ώψη της πώληση για με κάθε τρόπο. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει και τους ενεργητές οι οποίοι έχουν οποίοι πουλούν τα προϊόντα δικής παραγωγής αλλά και τους κυπουρούς θα ήθελα λοιπόν να ακούσω μια διευκρίνηση από την Κομισιόν για αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα. Ευχαριστώ Μάρκ. Τζορτ Ευχαριστώ. Να συγχαρώ τον συνάδελφό για την παρουσίαση. Το συγγνώμη που έχασα την παρουσίασή του σήμερα. Να αναφερθώ σε κάποια σημεία. Συμφωνώ με την πρόταση Κομισιόν για την απλούστευση του κανονισμού. Αν δείτε όμως το πολυάριθμο έγγραφα, τότε δεν πρόκειται καθόλου για απλούστευση. Πρόκειται για ένα ογκώδες έγγραφο και μία από τις ανησυχίες μας είναι ότι δεν θα γνωρίζουμε λεπτομέρειες μέχρι να δούμε την κατεξοδότηση πράξης ή τις εφαρμοστικές πράξεις ε, εκτελεστικές. Τώρα, η επάνηση της ε, βιομηχανίας του κλάδου φαίνεται πως είναι θετική, αλλά ένα σημείο θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το ζήτημα του κόστους. Βλέπω εδώ μια σειρά περιπτώσεων που υπάρχει δυνατότητα να καταλήξουμε σε υπερβολικό κόστος ε, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα προκαλέσουμε μεγαλύτερο κόστος ε, και αύξηση των ε, τιμών του τελικού προϊόντου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ του συναδέλφου που έλαβαν το λόγο. Να ακούσουμε τώρα την Κομισιόν. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Λάντισλαβ Μίκο από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ και μετά θα δώσω το λόγο στον Σέρτζο Σιλβέστρη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δυστυχώ ο αναπληρωτή Γενικό και κ. Ε, δεν είναι παρόν. Θα τον αναπληρώσω αν μου το επιτρέπετε για να απαντήσω στα, στους βουλευτές ε, που μίλησαν να ξεκινήσω λέγοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα πολύ τεχνικό φύσης, δύσκολο, καλύπτει πάρα πολλά φυτά, τα δημητριακά, τα ε, φρούτα, τα καλοπιστικά φυτά κλπ. Είναι λοιπόν περίπλοκος τομέας ε, με μεγάλη ποικιλία. Θέλησαμε όμως σε ένα έγγραφο να συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα θέματα, αλλά με κάποιες ιδιαιτερότητες κάποιες, ε, σε κάποιες περιπτώσεις. Θέλαμε λοιπόν να, να, να συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα είδη διότι θεωρούσαμε ότι εμπίπτουν στους ίδιους κανόνες. Το δεύτερο είναι ε, η τήρηση της βιοπικιλότητας. Η Γενική Διεύθυνση Υγείας Καταναλωτή αλλά και αυτής της Γεωργίας του περιβάλλοντος όλες λοιπόν οι γενικές διευθύνσεις ε, έχουμε κατά νου την τήρηση της βιοπικιλότητας, την ανάπτυξή της, την εξέλιξη και την προστασία της. Δεν ε, πρόκειται εδώ να για ε, μια προσπάθεια μείωση του αριθμού των σπόρων και των φυτών που υπάρχουν. Γνωρίζουμε την σημασία που πρέπει να αποδίδουμε σε αυτές τις ποικιλίε, ακόμα και αν δεν καλλιεργούνται σήμερα, διότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να βρούμε ε, γενετικές ποικιλίε και να χρειαστούμε να ξαναγυρίσουμε στις παλιές ε, παραδοσιακές ε, καλλιέργειες. Ε, μιλάω εδώ για αντοχή, για ανθεκτικότητα στις ασθένειες, την ανθεκτικότητα σε ξηρασία, στο ψύχος, όλες αυτές οι παλιές ποικιλίε μέσω της φυσικής επιλογής κατέδειξαν μια σειρά από ιδιότητες που θα πρέπει να προστατευτούν. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να θελήσουμε να πλήξουμε την βιοπικιλότητα. Για να απαντήσω σε κάποιες παρεμβάσεις, να πω πως ε, συμφωνούμε με τα συμπεράσματα του εισηγητή, κυρίου Σιλβέστρης, και συμφωνούμε με την δηλώσεις ε, κ. Ντόρφμαν και Κάπουλος Σάντος που έλεγαν ότι τα φυτά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα προτού να διατεθούν στην αγορά, ώστε αυτοί που αγοράζουν πρόκειται για επαγγελματία, γεωργό, έναν ε, δασοκόμο ή έναν ε, οποιοδήποτε πολίτη να μην μπορεί να εξαπατηθεί από εσφαλμένες ε, δηλώσεις ή βεβαιώσεις Αυτό το θέμα της πιστοποίησης έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία. Πάντως ε, έχουμε προβλέψει μια σειρά από απλουστεύσεις ε, για μια σειρά εμπλεκομένων δηλαδή προβλέψαμε κάποια κριτήρια φυσικά διότι θέλουμε να αποφύγουμε τις ε, αθέμητες ε, πρακτικές, ε, αλλά κριτήρια πολύ απλά για την καταγραφή των παραδοσιακών ποικιλιών, για κάποια βιολογικά φυτά και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα για τις ανταλλαγές μεταξύ ερασιτεχνών και εδώ απαντώ στον κύριο Ταραμπέλα, ή και για τα σπόρους που κρατάει στην αγρό του, στην αποθήκη του, ο, ο για να τους σπείρει την επόμενη χρονιά. Αν υπάρχουν ανταλλαγές ε, δωρεάν ανάμεσα σε εραστέχνες ή σε γεωργούς, ε, εκεί δεν προβλέπεται επιστοποίηση. θα πρέπει να διευκρινιστεί ενδεχομένως, αλλά δεν θελήσαμε. Μιλούσα χορήγηση δωρεάν ένας ε, γεωργός πολύ ε, σπόρους σε άλλο γεωργό, μιλάω για πώληση, τότε θα πρέπει να περνάμε μέσω του συστήματος πιστοποίηση. Αν δίνει όμως έτσι, δωρεάν, να χαρίζει σε κάποιους γείτονες, σε κάποιους φίλους ε, σπόρους, εδώ δεν απαιτείται την πιστοποίηση. Τώρα για να επανέλθω στις βιολογικές καλλιέργειες. Η βιολογική καλλιέργεια αφορά δύο είδη σπόρων. Σπόρων που βρίσκουμε στην αγορά για τη μεγάλη βιολογική καλλιέργεια, δηλαδή γεωργούς που φυτεύουν 50-100 εκτάρια σιτάρι και άλλα για την παραγωγή ψωμιού και τις ανταλλαγές με μικρούς, πολύ μικρούς ε, γεωργούς ή με εραστέχνες. Και εδώ υπάρχουν κάποιες διαφορές, ακόμα και αν τα πάντα καλύπτει η βιολογική γεωργία. Νομίζω ότι μεγάλες καλλιέργειες βιολογικές θα πρέπει να υπόκειται σε αυτήν την αρχή αλλά αν υπάρχει κάποια ευελιξία σε ζητήματα ποικιλιών ε, ε, μη συμβατικών. Έχουμε προβλέψει λοιπόν μια σειρά από παρεκκλήσεις διότι γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες της βιολογικής καλλιέργειας και θέλουμε να τηρηθούν. Ε, για τους εραστέχνες που ανταλλάσσουν βιολογικά, βιολογικούς πόρους και εδώ έχουμε προβλέψει ελάχιστες υποχρεώσεις. να απαντήσω σε όσους αναφέρθηκαν στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Έχουμε στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν πως αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές που όπως είπαν κάποιοι εξημών με ύψιλον ε, πολλούν και ζυζανιοκτώνα ε, καλύπτουν μόνο το 30% της αγοράς, δηλαδή 70% της αγοράς καλύπτεται από μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις ή ακόμα και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατανοούμε πως αυτές οι μικρές, πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να ε, τις πνίξουμε με μια σειρά από γραφειοκρατικές ε, ρυθμίσεις. Γνωρίζετε καλά διότι επειδή εξετάζεται και το πακέτο που φορά την υγεία των ζώων, των φυτών και τα φυτικών αναπαραγωγικού υλικού και ότι οι μικροεπιχειρήσεις θα εξαιρεθούν από την καταβολή ε, κάποιων τελών για, την, ε, για τους ελέγχους ε, που ενδεχομένως θα κληθούν να εφαρμόσουν. Αυτά, Πρόεδρε, σχετικά με τις απόψη μας φυσικά θα συνεργαστούμε με τον κύριο εισηγητή Σιλβέστρης αλλά και με την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ και να δώσω το λόγο στον Σέρτζο Σιλβέστρης για δύο λεπτά. Ναι, δύο λεπτά πάνω κάτω θα τα καταφέρεις. Ναι, αν χρειαστεί να πούμε περισσότερα, μπορούμε να το κάνουμε, να αναβάλουμε για την επόμενη εβδομάδα το επόμενο σημείο στη μερίζα που δεν είναι και το σημαντικό έτσι, να χρειαστούμε παραπάνω χρόνο. Αλλά θα είναι σύντομος Πρόεδρε. Ευχαριστώ του συναδέλφους για την ειλικρινή συζήτηση και για τον πλούτο των επιχειρημάτων. Σύντομα να αναφερθώ σε αυτά που σημείωσα με μεγάλη προσοχή και που θέλω σύντομα να σχολιάσω. Συμφωνώ με τον Ρότολφο συμμεριζόμαστε την ίδια προσέγγιση ως Αυτά που μόλι είπε η Κομισιόν μου φαίνονται σημαντικά. 30% τη αγορά βρίσκεται στις πολυεθνικέ που παράγουν και ζανιοκτώνα. Το 70 όμω εκπροσωπείται από μικρές. Και εγώ είμαι κατά τον τραστ. Το λέω ειλικρινά αυτό προς τον συνάδελφο Όσλινγκ. Γιατί αυτός που παράγει Ζανιοκτώνα και έχει μονοπόλιο, τότε ισχύει αυτό που ισχύει με, τα, με τους ιούς και τα αντιϊκά στην πληροφορική. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό το θέμα πολύ προσεκτικά, γιατί είναι αλήθεια ότι κανείς δεν θα πρέπει να έχει μονοπόλιο φυτικού υλικού και κατά συνέπεια του ελέγχου της παραγωγής και φυτοπαραγωγικής διαδικασίας και διατροφικής. Οπότε τους φόβους αυτούς τους συμμερίζομαι και τους λαμβάνω υπόψη μου σοβαρά. Συνάδελφος Κάντεμπαχ προέβαλε κάποια επιχειρημάτα τα οποία συμμερίζομαι ιδιαίτερα. Ξέρετε, στα μέρη μου υπάρχουν πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις και ελάχιστες μεγάλες η κληρονομιά τη βιοπικιλότητα είναι αυτό που χαρακτηρίζει την Ιταλική γεωργική παραγωγή. Μικρέ επιχειρήσει λοιπόν και βιωσιμότητα πάνε μαζί, είναι συμφασμένα. Για την απλούστευση και ο συναδελφό Ανιών και οι συναδελφοί Ρέιμερ έθεσαν το ίδιο θέμα. Δηλαδή, να περιοριστούμε σε ένα ενιαίο κανονισμό σημαίνει απλουστεύουμε ή αυτό παρουσιάζει τον κίνδυνο περαιτέρω περιπλοκότητας. Αυτό είναι αναπόφευκτο όμως. Το νέο κείμενο επιφέρει μειώσεις και στο αριθμό των οδηγιών αλλά και στο περιεχόμενο. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους μας. Ρόντους. Έθεσε διάφορα ζητήματα που διάθεση στην Κομισιόν. Να πω ταχύτατα ότι συμφωνώ πάνω με αυτά που είπε ο συνάδελφο Κάπουλα Σάντο. Δηλαδή σήμερα θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε δύο απαιτήσει σε δύο ανάγκες. Πρώτον, ότι αγοράζουμε αυτά που θεωρούμε ότι αγοράζουμε και πρέπει να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Δεύτερον, όποιο αγοράζει αυτό το υλικό, αυτό το υλικό πρέπει να είναι υγιέ. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν η βεβαιότητα ότι αγοράζουμε αυτό που θεωρούμε ότι αγοράζουμε μέσω συστήματο, δηλαδή πιστοποιήσεων που θα είναι σοβαρό και δεύτερον όποιος αγοράσει αυτό το υλικό όπω λέει προηγουμένω και ο Ντόρφμαν η ζημιά από ένα μη υγιέ προϊόν είναι τεράστια για μια γεωργική επιχείρηση γιατί είναι μια ζημιά που για να εκδηλωθεί χρειάζεται χρόνια και για να ξεπεραστεί χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια επενδύσεις και χρήση ζανιοκτώνων που προσβάλλουν τη γη. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να αποφευχθούν με ένα σύστημα πιστοποίησης και ελέγχων που θα αποτελεί εγγύηση για την βέλτιστη υγεία και κατάσταση του αγορασμένου υλικού. Και αυτό ακριβώς εννοώ το θα πρέπει να αγοράσουμε αυτό που θεωρούμε ότι αγοράζουμε. Ο κ. Σταραμπέλα στράφηκε προς την Κομισιόν η οποία ήδη απάντησε νομίζω Τώρα για, την, για τις ε, καταξιδότηση πράξεις είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε περιττέρω. Πάντως νομίζω ότι με αυτά τα πρώτα βήματα θα ξεκινήσουμε τη δουλειά μας, θα καταθέσουμε την έκθεση και θα αξιολογήσουμε και τις τροπολογίες που θα κατατεθούν, αλλά με πνεύμα απόλυτα επικοδομητικό και παρόμοιο με αυτό που καθοδήγησε τη σημερινή συζήτηση να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κάπουλα, τον Σκιώδη της εκθεσή μου και να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και ολόκληρη την Επιτροπή μας για τον χρόνο και την προσοχή που μου παραχωρήσατε. Και σήμερα, Πρόεδρε, απόλαυσα μεγάλη προσοχής από πολύ κόσμο που είχε συνδεθεί προηγουμένως στο streaming είδε να νόμιζε ότι θα έβλεπε τη συζήτηση για την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και αντίθετα είδε εμένα. Οπότε εποφολούμε λοιπόν και αυτή τη ευτυχού συγκυρία, 17 και ένα λεπτό, σταματάω να, σταματάω να μιλάω, μπορώ, ώστε να, να συζητήσουμε και να ψήφισουμε την, την ΚΑΠ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σέρτζο, να επιθυμήσω ότι στις 25 και 26 του Νοεμβρίου θα ξανασυζητήσουμε την έκθεση αυτή Προθεσμοί για την κατάθεση των τροπολογίων είναι η 4η Δεκέμβρη. Έχουμε λοιπόν χρόνο για να το εξετάσουμε το θέμα αυτό και να ανταπεξέλθουμε και να ανταποκριθούμε στις ευαισθησίες που εξέφρασαν οι συνάδελφοι. Προτείνω τώρα να σταματήσουμε για δύο λεπτά, να διακόψουμε μάλλον τις συνεδρίες για δύο λεπτά, ώστε να βρουν όλοι οι συνάδελφοι την ηλεκτρονική κάρτα ψηφορίας, γιατί χωρίς αυτήν σήμερα δεν γίνεται να ψηφίσετε με ανάταση της χείρας δεν γίνεται να ψηφίσουμε σήμερα. Βρείτε λοιπόν την κάρτα την ηλεκτρονική σας και σε δύο λεπτάκια ψηφίζουμε για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ένα λεπτό διάλειμμα. Είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να προχωρήσουμε, συνάδελφοι. Φτάσαμε σε μια στιγμή όπου βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, σε ένα σημείο δηλαδή το οποίο μας έχει απασχολήσει εδώ και πολύ καιρό. Πρέπει να δώσω λοιπόν το λόγο στους εισηγητές μας, θα πρέπει να τους ευχαριστήσω. Λουίς Κάπουλα Σκάντος, Τζοβάνι Λαβέκη, Ταντέν, Αλλά να ευχαριστήσω επίσης και όλη την ομάδα των διαπραγματεύσεων, όλους τους κοιόδης, όλους αυτούς που εργάστηκαν για αυτή την τόσο σημαντική σημερινή στιγμή. Νομίζω ότι θα πρέπει η Επιτροπή μας, Γεωργία και Ανάπτυξη Πέθρου, περήφανη για την δουλειά που έχει γίνει Νομίζω ότι δεν υπάρχει εμφωλία ότι ήμασταν στο ύψος της συναπόφασης που απορρέει από την συνθήκη της Λισαβόνας και μας δίνει τόσες αρμοδιότητες στη διαδικασία των αποφάσεων. Βεβαίως οι συνάδελφοί μας ενδεχομένω θα ήθελαν να πετύχουν περισσότερα, θα ήθελαν μια πιο θαραλέα ΚΑΠ, θα ήθελαν να πετύχουν κάτι παραπάνω ώστε να κάνουν πιο ανταγωνιστικούς, πιο ισχυρούς τους γεωργούς μας για να ανταποκριθούν σε ανάγκες που πηγαίνουν πέραν των προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο πλανήτης και χρειάζεται μια ισχυρή γεωργία. Αλλά το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων ήταν σημαντικό. Είχαμε πάνω από 50 τριμερείς ε, συναντήσεις με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Να ευχαριστήσω την Ιρλανδική Προεδρία του Σάμον Κοντ, τον Υπουργό και τη Λιθανική Προεδρία επίσης για το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής αυτή την διαπραγμάτευση. Τώρα, συναδελφοί, πριν να δώσουμε το λόγο στους τρεις ηγητές, θα πρέπει να κάνουμε μία δοκιμή, ένα τεστ, ώστε το σύστημα να είμαστε βέβαιοι ότι λειτουργεί. Σας παρακαλώ να βάλετε την ε, κάρτα και να ψηφίστε μόνο όσοι έχετε δικαίωμα και ενδεχομένω αυτοί που αντικαθιστούν. Να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφορία. Άρχεται η δοκιμαστική ψηφορία. Ψηφίστε δοκιμαστικά. Λειτουργούν όλα καλά, ρωτάει ο πρόεδρος. Έχουμε πάνω από μία, έχουμε μία παραπάνω ψήφο από τους μη γραμμένους. Έτσι. Ωραία. Τώρα ξεκινάμε με τους ηγητές. Σκάπουλα Σάντος, άμεσες πληρωμές και στήριξη της ανάπτυξης Πέθρου. Λουίς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα φτάνουμε σε μια φάση πολύ σημαντική αυτή τη τόσο μακροχρόνια διαδικασία στην οποία αφιερώσαμε πολλέ ώρε εργασίας, όπου συμμετείχαν πάρα πολλοί μέλη τη επιτροπή μα, τα μέλη των και υπάλληλων γραφείων μας, οι εκπρόσωποι των φορέων των γεωργών που συμμετείχαν στις επαφές που είχαμε στις διάφορες χώρες κλπ. κλπ. Συμμετείχε λοιπόν πάρα πολλοί κόσμο σε αυτή τη δικασία και είμαστε πολύ περήφανοι για τη δουλειά που έχει γίνει επειδή επιπλέον θεωρούμε ότι έχουμε κάνει το καθήκον μας και χαίρομαι που είμαι σε θέση να πω στους Γεωργούς ότι από το 2014 θα έχουμε μια καλύτερη ΚΑΠ χάρη ακριβώς στην δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις συνεργίες του η μελλοντική ΚΑΠ θα περιλαμβάνει μεγαλύτερη δικαιοσύνη και ισότητα μεταξύ των γεωργών και των χωρομελών. Θα έχουμε επίση και περισσότερο ρόλο του περιβάλλοντο. Θα σεβόμαστε περισσότερο το περιβάλλον, κάτι το οποίο ανταποκρίνεται βεβαίω και στι επιθυμίε όχι μόνο των γεωργών αλλά και των καταναλωτών. Επίση θα έχουμε μια μεταρρύθμιση απλουστευμένη, πιο απλή. Δεν ενδεχομένως είναι η επιθυμητή ή η ιδανική μεταρρύθμιση, αλλά είναι η μεταρρύθμιση για την οποία υπήρξε συνένεση. Χρειάστηκε να γίνουν παραχωρήσει, όμω νομίζω ότι είχαμε και επιτεύγματα. Και το τελευταίο επιτεύγμα και επιτυχία ήταν να πετύχουμε από το Συμβούλιο να τηρήσει την συνθήκη τη Αβώνα και είπαμε εμεί ότι δεν θα κλείσουμε την διαπραγμάτευση μέχρι όλα τα θέματα τα οποία ήταν υποδιαπραγμάτευση να συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να επιβάλλουμε στο Συμβούλιο μία αλλαγή εντολής ώστε να είναι παρόντες στην συζήτηση όλων των θεμάτων. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο. Στο μέλλον θα πρέπει να υιοθετήσουμε σημαντικές αποφάσεις, ξεκινώντας από τη σημερινή ψηφοφορία, και την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν επειδή υπήρξε μια πιστή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων και θεωρώ ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια, όχι μήνες, χρόνια, χρόνια δουλειά έχει λειτουργήσει σωστά η συνεργασία μεταξύ των πολιτικών ομάδων και νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι το καλύτερο ως καρπός που έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Ο Μισελ Τατέν για την κοινή ΚΟΑ. Μισελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους και οδησηγητές, ε, τη γραμματεία βεβαίως, το επιτελείο που με βοήθησε. Όλους αυτούς που μας βοήθησαν για να ετοιμάσουμε για πρώτη φορά ένα νομοθέτημα από τη συναπόφαση στη Γεωργία. Με μεγάλη προσοχή, φρόνηση και ευφυΐα και με μια πολύ θετική Προεδρία, την Ισλανδική, με μια επιτροπή που είχε την πρόθεση και διάθεση να προχωρήσει και να προωθήσει τα ζητήματα στις γραμμές της ε, πολιτικής της γεωργίας. Σημειώνονται πιστεύω σημαντικές πρόοδοι, ε, ιδιαίτερα η πρόοδο στους τομείς του, αμπε, του αμπελοϊνικού ε, και πευτικών. Δυστυχώς δεν έχουμε προχωρήσει επαρκώς στον χώρο του γάλακτο, στον τομέα του Γάλακτο. και λυπούμε ιδιαίτερα γιατί φοβούμε ότι με τα υφιστάμενα νομοθετήματα δεν είναι ασφαλή, ο τομέα, κινδυνεύει. Η πρόοδο ω προ οργανώσει των παραγωγών έχει νομική βέβαια σημασία και αξία, παραμένει όμω ένα μέσον και όχι μια συνταγή. Άρα ο κάθε γεωργός στην κάθε χώρα μέσω των ε, νομοθετικών ε, ε, μέσων που θα έχουν σε θέση του ανάλογα με το κράτο θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Από κοινού πιστεύω καταφέρουμε να χτίσουμε μια ΚΑΠ πιο δίκαιη, πιο σωστή αλλά και πιο δυναμική πιστεύω. Δεν θα αποφασίζονται τα πάντα από τις Βρυξέλλες θα μπορούμε χάρη στην πολιτική αυτή να αφήσουμε τις επιλογές στον ίδιο τον παραγωγό, στον ίδιο τον φορέα, τον παράγοντα, στην κάθε περιοχή για να δοθούν αποτελέσματα ουσιαστικά. Εάν θέλουμε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για την υλοποίησή της βεβαίως και πάλι ευχαριστώ όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου. Πιστεύω ότι χάρη, ότι μέρος αυτής της μεταρρύθμισης τους ανήκει. E και τώρα το λόγο έχει ο Τζοβάνι Λαβία για τη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΑΠ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνεργάστηκαν σε αυτή τη μακρά διαδικασία που ξεκίνησε στις 12 Οκτωβρίου του 2011 με την παρουσίαση της πρότασης πλευράς ε, κομισιών και τώρα δύο χρόνια σχεδόν αργότερα μας οδηγεί στο να ολοκληρώσουμε μια περίπλοκη μεταρρύθμιση στην πλέον περίπλοκη στην ιστορία της ΚΑΠ. Για πρώτη φορά βρισκόμαστε με έναν προπολογισμό χαμηλότερο από τον προηγούμενο και δώσαμε έναν αγώνα τόσο με τα άλλα θεσμικά όργανα ε, μια αντιπαράθεση προκειμένου να βελτιωθεί η μεταρρύθμιση της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής αλλά ιδιαίτερα και σε επίπεδο οικονομικών πόρων, διότι αυτή η πολιτική θα έπρεπε τα προσεχή έτη να μπορέσει να έχει μια πρικοδότηση κατάλληλη ή ικανή προκειμένου να θεωρηθεί ως η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική, μια πολιτική ικανή να δώσει απαντήσεις όχι μόνο στις ανάγκες των γεωργών αλλά και στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Δεσμευθήκανε ώστε η αρχική πρόταση να μπορέσει να βελτιωθεί και έτσι να έχουμε μια κοινή αγροτική πολιτική πιο εύκολη στην εφαρμογή της. Λιγότερο περίπλοκη για τους γεωργούς και νομίζω ότι προς την κατεύθυνση αυτή πολλά πετύχαμε, αλλά δράσαμε και όλοι μαζί, όλες οι πολιτικές ομάδες, ε, έτσι ώστε να υπάρξει Έλεγχο των Ευρωπαίων πολιτών επί τη πολιτική αυτή και ό,τι κάναμε για την ευθυγράμμιση με τη Συνθήκη Λισαβόνα πηγαίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Διότι και η γεωρική πολιτική θα πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά από τι ε, κυβερνήσει, αλλά θα πρέπει να διαδραματίζει για το Κοινοβούλιο ένα σημαντικό ρόλο και θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι καλό αποτέλεσμα, σίγουρα καλύτερο από την αρχική πρόταση. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Τζοβάνι. Και τώρα, στην άλλη ξεκινάμε με τις ψηφοφορίες. Όπως είπα στην αρχή, θα έχουμε τέσσερις ψηφοφορίες. Μία ψηφοφορία για κάθε φάκελο, για κάθε θέμα. Οι ψηφοφορίες θα είναι χωριστές, αλλά σε περίπτωση που δεν κατορθώσουμε να πετύχουμε την ε, να πετύχουμε συμφωνία, σε έναν από τους τέσσερις φακέλους, τότε όλη η διαδικασία της ε, μεταρρύθμισης καταπίπτει. Ξεκινάμε με την ψηφοφορία σχετικά με τις άμεσες πτωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ψηφίζουμε. Dichiaro chiusa la votazione του ψηφορία. Εγκρίθηκε 31 ψήφοι υπέρ, 8 ψήφοι κατά και 2 εποχέ. Τώρα ψηφίζουμε επί του δεύτερου φακέλου. Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων. Κανονισμό ενία ΚΟΑ. Άρχιτη ψηφοφορία. Chiusa la votazione. Πέρα Εγκρίθηκε 27 ψήφοι υπέρ, 14 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Και τώρα περνάμε στην ψήφιση του τρίτου φακέλου. Στήριξη της αγροτική ανάπτυξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο. Αγροτική ανάπτυξη. Άρχιτη ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. ...35 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, 3 αποχές. Εγκρίθηκε και ο τρίτος φάκελος. Και τώρα ψηφίζουμε το τελευταίο φάκελο που αφορά στη χρηματοδότηση, διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινή αγροτικής πολιτικής. Άρχη ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε και ο τέλος φάκελος, 35 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, καμία αποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να συγχαρούμε τους τρεις συζητητές μας. Έχουμε ε, την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που μόλις εγκρίθηκε. Grazie, grazie a ε, ε, tutti i colleghi. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και θα έλεγα πως τώρα μπορούμε να περάσουμε στα μεταβατικές, μεταβατικές διατάξεις ένα άλλο σημαντικό θέμα παρακαλώ τους συναδέλφους να δώσουν την δέουσα σημασία. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή, στον Άλμπερτ Ντές Πολλές οι τροπολογίες που κατέθεσαν αφορούν το ζήτημα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ που μόλις εγκρίναμε. Θεωρώ πως είναι σημαντικό ο Άλμπερτ να μας ε, αναφέρει πρωτού περάσουμε στις ψηφοφορίες ε, τις εργασίες του, την εργασία του και μετά θα περάσουμε, να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Άλμπερτ Ντέσσα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, και ολοκληρώθηκε τώρα μεταρρύθμιση και τη ευρωπαϊκή πολιτική, πρέπει να συμφωνήσουμε για τι μεταβατικέ διατάξει. Έτσι ώστε να συνεχιστεί, η... να παραμείνει δηλαδή ενισχύει ο κανονισμό, μέχρι ότου αρχίσει να εφαρμόζεται ο νέο κανονισμό, η νέα κοινή γεωργική πολιτική. Η δική μου έκθεση στόχο έχει να προσπαθήσουμε να ε, διατηρήσουμε στο δεύτερο πυλώνα τα προγράμματα, εδώ διαφοροποιούμαστε σε σχέση με την πρώτη ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θέλουμε για τους γεωργούς και το 2014 να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ε, βεβαιότητα για το τι θα συμβεί. Τεχνικού χαρακτήρα έκθεσή μου, διαφορές μεταξύ των πολιτικών ομάδων δεν εμφανίζονται, γενικά επικρατεί ομοφωνία. Θα ήθελα να ευχαριστώ τους συναδέλφους γιατί ήταν μεγάλη η χρονική πίεση και εργαστήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρετε πόσο ολοκληρώνονται τα θέματα της γεωργικής πολιτικής και εδώ στο Κοινοβούλιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συνεργάτες και τις συνεργάτητες και τους σκιώδεις, σκιώδεις με τους οποίους συνεργαστήκαμε και μπορούσαμε να βρούμε μια κοινή γραμμή. Θα παρακαλώ τον Πρόεδρο να μου δώσει το λόγο ε, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας πριν ε, από τις ψηφοφορίες για τις τροπολογίες 66, 75 και 23, 66, 75 και 23, γιατί θέλω να κάνω προφορικές προτάσεις τροπολογίας. Νομίζω ότι χάρη στην πρόταση αυτή μπορούμε να βρούμε τις κατάλληλες, τις αρμόνισες μεταβατικές διατάξεις για την ε, γεωργία της Ευρώπης, έτσι ώστε αυτή να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και σε όρους ασφάλειας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Άλμπερτ. Ο Άνδριος ζήτησε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση πολύ σημαντική για την ε, μεταβατικές διατάξεις. Θα ήθελα να επίσω την προσοχή του σώματος ε, την τροπολογική τροπολογία 23 που έχει κατατεθεί και μιλώ ως ε, σκιώδης ηγετής, η τροπολογία αυτή είναι απαράδεκτη διότι προτείνεται να μεταφερθεί το ζήτημα του πρασινίσματος. Το είχαμε θίξει καρδιά τη τις συνεδρίαση, αλλά θα ήθελα να το υπενθυμίσω και εδώ. Δεν μπορούμε λοιπόν όπως έχουν τα πράγματα να δεχθούμε αυτή την τροπολογία διότι ε, θεωρείται απαράδεκτο υπό ε, τη μορφή που μας έχει παρουσιαστεί. Θα ήθελα επίσης να εκφέρω την ίδια άποψη για την τροπολογία 107 που κατά την άποψή μου είναι απαράδεκτη διότι κατά, σύμφωνα με αυτή ε, προβληματική αφορά ζήτημα της διαφάνειας και ως εκ τούτου η τροπολογία αυτή θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ζητήσουμε την απόσυρση των δύο αυτών τροπολογιών όσο έχουν και έτσι να μην ψηφιστούν από την Επιτροπή. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικά, ε, σημαντικές αυτές οι τροπολογίες και ήθελα να το αναφέρω πριν να περάσουμε στην ψηφοφορία. Λοιπόν, συνάδελφοι, ο Έρικ, μάλλον Έρικ, μόλις ψηφίσαμε ε, τέσσερα ε, θέματα που αφορούσαν την μετάρρυθμιση. Δεν υπάρχει, μάλλον η σύνδεση είναι πολύ ουσιαστική με το έγγραφο του Άλμπερτ για τις μεταβατικές διατάξεις, αλλά δεν υπάρχει κάποια διαδικαστική διαδικασία που να εμποδίζει στις μεταβατικές διατάξεις να, παρε, να να παρέμβουν σε αυτά που ψηφίσαμε. Λοιπόν, θα ζητήσουμε εμείς τη ψηφοφορία και με την ψηφοφορία θα λάβουμε υπόψη φυσικά τις ευαισθησίες που μόλις μας εξέφρασες. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις θα δώσω το λόγο στις διαδικασίες ψηφοφορίας. Παρακαλώ, έχεις το λόγο Μάρτιν. Θα ήθελα απλώ να υποστηρίξω το αίτημα του κύριου Άντριου. Γιατί αν ψηφιστεί αυτό, τότε το πρασίνισμα, η έκθεση για το πρασίνισμα πάει για το 2016 αντί να τεθεί σε ισχύ όπως προβλέπει το 2015, δηλαδή όπω ψηφίσαμε με την προηγούμενη έκθεση για την κοινή ιδιορκή πολιτική. Άρα αντιφάσκουμε. Αν δηλαδή ψηφίσουμε την 23 και την 37, εν τέλει θα πρέπει να στραφούμε κατά των μεταβατικών διατάξεων για να είμαστε συνεπεί με την Κουγουπού. Α είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Ο Άλμπερτ Ντέσσα, αν έχει την καλοσύνη, να αποσύρει τις τροπολογίες του. Ιδάλω θα πρέπει να καταψηφίσουμε τι μεταβατικέ διατάξει για να είμαστε συνεπείς με τα όσα μόλις ψηφίσαμε για τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής πολιτικής και με αυτά που μας ζητάτε να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι θα πρέπει να γνωρίζουν τι ακριβώς ε, θα ψηφίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν επιφυλάσσομαι να δώσω το λόγο από τις τοπολογίες αυτής των συνάδελφο και φυσικά να προσέχουμε τι ψηφίζουμε ώστε η στάση μας να μην είναι αντιφατική από διαδικαστικής πλευράς εμείς θα πρέπει να ψηφίσουμε. Ελπίζω η Επιτροπή Γεωργίας να δείξει συνέπεια και συνοχή. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 4 του εισηγητή. Άρχιτε ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα ψηφοφορία. Δεκτή. Περνάμε στην τροπολογία τη συμβαστική υπαριθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Επί της τροπολογίας 1. Συμβαστική. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Και τώρα περνάμε στην συμβαστική τροπολογία υπερθμών 2. Άρχιτη ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. προσέξτε γιατί υπάρχει ένα λάθος στον κατάλογο. Περνάμε στη τροπολογία 62. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 62. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 65. Ο Λενίτσακ. Άρχιτε ψηφοφορία. Επί της 65. Έληξη ψηφοφορία. Τώρα περνάμε στην 66 και δίνω το λόγο στον συνάδελφο Ντες, Άλμπερτ. Έχεις το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στις τροπολογίες αυτές, την 66, Μαρκίνες, 68 Κέστιγκερ και 69, Αντρέ, υπάρχουν ε, διαφορετικές πληροφορίες. Δεν θέλω συγκεκριμένε ρωτήσεις να υποβάλω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταλάβω. Εάν ψηφίσουμε αυτές τις, ψηφοφο... τις ε, τροπολογίες, θα έχουν επιρροή ως προς τις εθνικές ε, ως προς την κάλυψη εθνικό επίπεδο, εάν εγκριθούν αυτές οι τροπολογίες, τα ποσά που την στην εθνική κατανομή θα επηρεαστούν, αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας απαντήσει. Ο Άλμπερτ έθεσε ερώτημα προς την Κομισιόν. Η Κομισιόν είναι παρούσα. Όχι. Παρακαλώ, ο λόγος στην Κομισιόν, αν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα του συνάδελφου Ντέσσερ. Ευχαριστώ. Στη θέση του κυρίου Νία ονομάζομαι Κριστίνα Μπόκμαν. Φυσικά για τα ανώτατα όρια. Τα ανώτατα όρια είναι αυτά που έπρεπε να είναι, όπως αναφέρονται στο παράρτημα. Λοιπόν, δεν πρόκειται να επηρεαστούν άρα τα ποσά ανακράτους μέλος. Τα ποσά έχουν ως έχουν στο παράρτημα του κανονισμού. Ωραία, ευχαριστούμε την Κομισιόν. Και μπορούμε να περάσουμε ψηφοφορία επί του άρθρου 66. Άρχεται ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Chiusa la votazione. Πέρα ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 67 της συναδέλφου Λούλινγκ. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίζουμε επί της 67. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 68. Άρχιτη ψηφοφορία. Έληξε, όχι. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτή. Τροπολογία ΣΕΤΕ του εισηγητή. Ψηφίζουμε επί της 7. Ψήφισαν όλοι. Έληξε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 69 Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Έληξε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 70. Ψηφίζουμε επί της 70. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε επί της 71. 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. Τροπολογία 8 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Έληξη ψηφοφορία εγκρίνεται. Και τώρα 73. Ψηφίζουμε πέρα ψηφοφορία. Δεκτή. Τοπολογία 74. Αρχίζει ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτή 74. Και τώρα έχουμε την προφορική τροπολογία του εισηγητή. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο Άλμπερτ Ντες. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Προκύπτει απαραίτητη αυτή η τροπολογία και παρακαλώ τους συναδέλφους να με υποστηρίξουν. Δεν επηρεάζει την κατανομή των κονδύλων μεταξύ κρατών μελών. Εδώ Απλώς τα κράτη-μέλη διατηρούν τη δυνατότητα για την έγκριση των ε, συνδεδεμένων ανισχύσεων μετά την έγκριση της Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό για ορισμένα κράτη-μέλη και θα ήθελα να το υποστηρίξετε. Συνεχίζουμε με την Ψηφίζουμε. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτή. Συμβαστική τροπολογία υπερθμών 3. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Έληξε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 του Σιγητή. Άρχιτη ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. Δεκτή. 90 τροπολογία. Ψηφίζουμε επί της 90. Άρχιτη η ψηφορία. Ο Άγνιος, ζήτησε το λόγο. Πρόεδρε, βλέπω ότι θα προκύψει κατά πόσο πιθανότητα προφορική τροπολογία. Έτσι είναι. Ναι, Ορθό. Ορθό. Είστε κατά αν υπάρξει ε, ονομαστική ψηφοφορία, είμαι κατά ονομαστική ψηφοφορία. Τη Συγγνώμη, τη τη τροπολογίας. Κατά τη ονομαστική της προφορικής τροπολογίας. Συγγνώμη. Εντάξει, θα, θα το ιδιωθώσουμε, θα ψηφίζουμε δίχως την ε, προφορική τροπολογία. Ο Λουί έχει το λόγο. Ναι, πρόεδρε. Θα ήθελα να πιστώ την προσοχή πως ε, πρόκειται για μια τροποποίηση που δεν τροποποιούσε την ουσία της τροπολογής. Θα θέλαμε να βάλουμε την ίδια ημερομηνία που περιλαμβάνεται στο σχετικό εκτιμώντας. Οι νομικές επιπτώσεις θα είναι οι αυτές. Ε, πρόκειται για μια τροπολογία διευκρινιστική του νομοθετικού κειμένου, αλλά οι επιπτώσεις θα είναι οι αυτές. Δεν πρόκειται να αλλάξει η ουσία Εν σύμφωνα με τον κανονισμό, εάν έχουμε μία ένσταση, τότε η τροπολογία παραμένει ως έχει, εκτός αν έχετε πείσει τον κύριο Άγνιο. Δεν νομίζω ότι οτιδήποτε και να πει κάποιος εδώ θα με πείσει. Ευχαριστώ. Σαφέστατο αυτό που είπατε. Λοιπόν, ψηφίζουμε επί τροπολογία 90 χωρίς αυτή τη διόρθωση της, της προφορικής τροπολογίας. Άρχιτε η ψηφοφορία. Έλεξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 91. Άρχιτε η ψηφοφορία. Πέρασε εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Έληξε η ψηφοφορία. Δεκτή. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία υπαρθμών 23 του εισηγητή και θα δώσω το λόγο στον Άλμπερτ Ντες. Άλμπερτ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα αυτό, μια σύντομη εξήγηση. Στόχος της τροπολογίας είναι ο τελευταίος στόχος θα ήταν με αυτή την τροπολογία να αμφισβητηθούν οι ε, μεταρρυθμίσεις της ε, κινησιορικής πολιτικής. Έχω μιλήσει με, την νομική, με τους νομικούς πραγματογνώμονες και επειδή είναι περίπλοκο το ζήτημα και για τα κράτη-μέλη και επειδή διαπιστώθηκε ότι ορισμένα ζητήματα, για να σας υπενθυμίσω, ε, ε, ήταν πολύ δύσκολο να τηρηθούν οι διατάξεις για τα κράτη-μέλη, προτείνω για τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34 εφαρμογή όχι από το 2016 αλλά το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου του 2016 έτσι ώστε να μην έχουν κανένα εμπόδιο στην εισαγωγή αυτών των διατάξεων ενωρίτερα, εάν το επιθυμούν, τα κράτη-μέλη. Ξέρω ότι πολλά πράγματα ε, αναφέρεται ότι πρέπει να μετα πρέπει να αναθεωρούνται σε επίπεδο Βρυξελών και πολλά, πολλές από τις δετάξεις αρχίσουν να εφαρμόζονται από το 2015. Αυτό όμως με παράλληλο το πρασίτισμα στον πρωτοπυλώνα, θα μας προξενήσει πολλές δυσκολίες. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν που δεν η πρόθεσή μου να αφισβητήσω η αδίποτε μεταρρύθμιση. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα, τεχνικά δυνατό ζήτημα. Λέμε λοιπόν το αργότερο, το 2016, πρέπει να τεθούν τα πάντα σε εφαρμογή έτσι ώστε να έχουμε την ταχύτερη δυνατή εισαγωγή, υλοποίηση αλλά και χωρίς να παραβλάπτουμε οποιαδήποτε πρόθεση ή δυνατότητα παρέκτηση κάποιο το για ταχύτερη εισαγωγή, αν το επιθυμεί αυτό διατάξω. Αυτή είναι η παράκλησή μου και η τροπολογία. Ευχαριστώ. Βρισκόμαστε σε διαδικασία συναπόφασης. Αυτή είναι η πρώτη πράξη μετά θα πέρασε το Συμβούλιο, μετά συζητήσεις. Θα ήθελα να καθησυχάσω όλους ε, όσοι εξέφρασαν ανησυχίες. Λοιπόν, περνάμε στις ψηφοφορίες. Άρθρο, τροπολογία 23, η ψηφοφορία. Chiusa la votazione. Έληξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ε, τώρα μπορούμε να περάσουμε στην τροπολογία 103. Ψηφίζουμε την 103. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. Δεκτή. 105 τροπολογία. Ψηφίζουμε. Έληξη ψηφοφορία. 106. Άρχη ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίνεται. 107. Τροπολογία 107. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 21 υπέρ, 18 κατά. Τροπολογία 108. Ψηφίζουμε. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτή. 109. Ψηφίζουμε επί της 109. Έληξε. Δεκτή. Συμβαστική 5. Άρχιτη ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 29 του εισηγητή άρχιτη ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. Τροπολογία 30 του εισηγητή. Έληξη ψηφορία. Δεκτή. Τροπολογία 31. Άρχιτη ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίνεται. 110. Άργεται Πέρας. Δεκτή. 113. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Άρχεται. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 114. Άρχεται η ψηφοφορία. Έλλειψη. Δεκτή. 33 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφορία. Έληξε. Δεκτή. Ψηφίζουμε επί της 34. Ψήφισαν άπαντες. Έλικρη ψηφοφορία. Δεκτή. Και τώρα συνάδελφοι θα πρέπει να ψηφίσουμε επί του ψηφίσματος νομοθετικού περιεχομένου όπως τροποποιήθηκε. Ψήφισαν όλοι. έγινε δεκτή με συντριπτική πλειοσοφία, 35 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά. Και τώρα ψηφίζουμε την απόφαση έναρξης ε, διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. άρχιτη ψηφοφορία. Έληξε. εγκρίνεται με συντηρητική πλειοψηφία. Θα πρέπει να εκφράσουμε την γνώμη μας για τη σύνθεση της ε, διαπραγματευτικής ομάδας. Άρχη ψηφοφορία, λήξη ψηφοφορίας. Και αυτό έγινε δεκτό. Προτού να περάσουμε στο τελευταίο σημείο της σήμερων, θα ήθελα εξ ονόματος όλων να χαιρετήσω ένα συνάδελφο που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα αλλά ψήφισε κατά τη διάρκεια των Ολομέλειας του Στρασβούργου. Ο συνάδελφος Πάπα Στάμκος θα ήθελα εξ ονόματος όλων μας να του στείλουμε ένα θερμό χαιρετισμό διότι ήταν πρωταγωνιστής αυτής της μεταρρύθμισης δυστυχώς δεν βρίσκεται μαζί μας και του ευχόμαστε να επιστρέψει ανάμεσά μας το συντομότερο. Ε, το σημείο 12 στη μέση διατάξη είναι πολύ γρήγορο. Πρόκειται σε αγροτικές και αλευτικές σταριστικές. στην ακίνηνο τεχνικής φύσης υπάρχει μία και μοναδική ψηφοφορία, μια και έξω. Αν συμφωνείτε θα την κάνουμε ευθύς αμέσως ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό μπορούμε να περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημέρας. Ευχαριστώ όλους τους αδέλφους. Παρουσίαση εξ ονόματος ε, της Επιτροπής σχετικά με την ομάδα υψηλού επίπεδου για τα δικαιώματα φύτευσης αμπελώνων. Είχαμε ζητήσει ε, μέρους όλων των συντονιστών η Κομισιόν να μας ενημερώσει σχετικά με την πρόοδο στην ομάδα υψηλού επίπεδου, μόνο ότι η μεταρρύθμιση που μόλις έχει εγκριθεί έδευσε κάποιες ενδείξεις, αλλά δεδομένου του ότι εγκρίθηκε από την συνεδρίαση των συντονιστών, βρίσκεται στη μέση ένταξη και αν οι συνάδελφοι που δεν ενδιαφέρονται εγκαταλείψουν την αίθουσα, θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν Τζορίλα από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Yes, Just to listen if there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 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχει τελειώσει το διάλειμμα, δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής τώρα και ελπίζω, ελπίζω να μας αφήσετε σε ησυχία να συζητήσουμε με την Επιτροπή για να τον ακούσουν και οι συνάδελφοι ως αρμόζε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω ότι η ομάδα υψηλού επίπεδου για τα δικαιώματα φύτευσης δημιουργήθηκε από τον Επιτροπό Τσόλο το 2012 μετά από την θέση πολλών χωρών μελών και του Κοινοβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα φύτευσης. Τα χειρότερα θέματα συζήτησης της ομάδας υψηλού επίπεδου που συνήλθε το 2012 ήταν τα εξή. Η λειτουργία του μεταβατικού καθεστώτος δικαιωμάτων φύτευση σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό για, κάθε, για κάποιες χώρες μέλη κατέδειξε το περιορισμό του συστήματος αυτό δικαιωμάτων φύτευσης όσον αφορά την άπτυξη ενός ανταγωνιστικού τομέα. Κατέδειξε επίσης και μια μεγάλη απόκληση όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των συστημάτων από χώρα σε χώρα. Και μάλιστα στην ίδια χώρα και σε περιφερειακό επίπεδο, κάτι το οποίο οδηγεί σε στρεβλώσεις στην κοινότητα. Η ομάδα μελέτησε επίσης και, το, και την πιθανή επίπτωση του τέλους του δικαιωμάτων φύτευσης και για τον κλάδο αλλά και για την αγορά. Παρόλο που το Ευρωκοινοβούλιο και, κάθε, και κάποιες χώρες μέλη και κάποιοι επαγγελματικοί, επαγγελματικές οργανώσεις επιθυμούν την, την διατήρηση του τωρινού συστήματος, υπάρχει μια ευρεία συνένεση μεταξύ οργανισμών και χωρών μελών για ένα νέο σύστημα που αφορά την επέκταση των δικαιωμάτων φύτευσης που θα είναι πιο ευέλικτο και που θα βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα εξή σημεία διαχείριση από τις δημόσιες αρχές για όλες τις κατηγορίες, τις κατηγορίες ε, νέων δικαιωμάτων φύτευσης, έκδοση νέων αδειών για νέες φυτεύσεις στο επίπεδο του 1% της επιφάνειας των αμπελώνων ευελιξία των χορμελών όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τις γεωγραφικές ενδείξεις με τη δυνατότητα να μειώσουν την ανάπτυξη σε κάτω από 1%. Ο στόχος εδώ είναι να επιτρέψουμε την ανάπτυξη του κλάδου όμως με μια ρήτρα, με μια δικλίδα ασφαλείας ώστε να μην έχουμε δυσανάλογη ανάπτυξη. Η ομάδα επίσης υψηλού επίπεδου προβλέπει και την ανάγκη διαβούλευσης με επαγγελματικούς, με επαγγελματικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τις φορές του κλάδου για την ρύθμιση των νέων φυτεύσεων ιδιαίτερα σαν αφορά τους ίνους ε, γεωγραφικής, ε, προέλευσης αλλά και για τους υπόλοιπους ίνους. Η συνένεση που επιτεύχθηκε στο Τέλο τη θητεία τη ομάδα ψηλού τέλη Δεκέμβρη 2012, αντανακλάται νομίζω σωστά στην θέση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για ένα αναλλακτικό σύστημα στο μεταβατικό καθεστώς. Υπήρξε πολιτική συμφωνία, επιβεβαιώθηκε εδώ σήμερα και όπω ξέρετε το νέο σύστημα αδειοδοτήσεων θα τεθεί σε ισχύ το 2016 και θα πηγαίνουμε στο 2030. Θα υπάρξει και ενδιάμεση αναθεώρηση στα μέσα αυτής της περίοδου όλου του συστήματος. Πρόεδρε με την άδεια σας να υποφεληθώ της ευκαιρίας για να απευθύνω μια, μάλλον για να θίξω μια προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν της κυρίας Λούλιν και του κυρίου Ντεκάστρο εξ ονόματος Επιτροπής ε, Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου του Κοινοβουλίου. Η ερώτηση, οι ερωτήσεις Λούλιν Ντεκάστρο αφορούν το μέλλον του κλάδου του Ίνου και τις προθέσεις της Κομισιόν. Καταρχάς, να επαναλάβω, επιτρέψτε μου, όπως κάναμε και στην έκθεση του 12 που στείλαμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ότι έχουμε μια θετική αξιολόγηση όσον αφορά την αθεώρηση του κλάδου των ίνων. Κάποια μέτρα εξαφανίστηκαν χωρίς ο κλάδος να αντιμετωπίσει προβλήματα. Έχουμε και νέα μέτρα, ιδιαίτερα τα εθνικά προγράμματα υποστήριξης, τα οποία θεσπίστηκαν με τρόπο ευέλικτο και πολύ αποτελεσματικό. να επιμείνω ότι για τον τομέα του ίνου να πω ιδιαίτερα ότι η Κομισιόν δεν έχει καμία πρόθεση να αναθεωρήσει ή να μεταρρυθμίσει έναν κλάδο ο οποίος μόλις τώρα πρόσφατα ήταν αντικείμενο μεταρρύθμισης. Το λέω αυτό στην επιστολή ως απάντηση στο ερώτημα αν η Κομισιόν έχει πρόθεση μεταρρύθμιση στο κλάδο αυτό. Όχι, η Κομισιόν έχει καμιά πρόθεση μεταρρύθμιση σε αυτόν τον κλάδο. Όπως γνωρίζετε, η μεταρρύθμιση που θα υιοθετηθεί πιθανότατα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις ερχόμενες εβδομάδες ήδη προβλέπει κάποια νέα εργαλεία τα οποία είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στον αμπελοϊνικό τομέα και ιδιαίτερα όσον αφορά τα προγράμματα υποστήριξης προς τον αμπελοϊνικό τομέα ώστε να θεσπιστούν νέα μέτρα, ιδιαίτερα όσον αφορά την προώθηση στις εσωτερικές αγορές, ώστε να καλύπτεται και το θέμα της καινοτομίας. Τα δύο αυτά μέτρα, τα μελλοντικά προγράμματα μπορούν να τα υιοθετούν, κατά το οποίο θα διευκολύνει όλη την προσπάθειά μας της μεταρρύθμισης ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Αυτά τα προγράμματα συμβάλλουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τα διαφορετικά μέτρα όπως η αναδιάρθρωση, οι επενδύσεις, η καινοτομία, η προώθηση και αυτά θα συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα, όπως έλεγα. Να προσθέσω τέλος ότι μετά από τη συζήτηση που είχαμε στο ΟΗΒ σχετικά με κάποια προϊόντα του κλάδου του ίνου με χαμηλή περιοκτικότητα σε αλκοόλ θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας και με το Συμβούλιο τη δημιουργία θέσπισης ευρωπαϊκών κανόνων για αυτό το τμήμα της αγοράς για τα μερικώς μη αλκοολούχα ποτά για τα οποία δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βλέπουμε ότι αυτό οδηγεί σε μια στρέβλωση στην εσωτερική αγορά. Αυτό το αναφέρω ως μελλοντική σκέψη για ένα θέμα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Επιμένω όμως ότι η Κομισιόν δεν έχει πρόθεση μεταρρύθμισης της μεταρρύθμισης, αλλά αντίθετα θέλει να την δρομολογήσει, γιατί θέλουμε ήδη από το 2014 τα νέα μέτρα να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα υποστήριξη των αμπελώνων της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συγγνώμη για την παρουσίασή σας. Μήπως έχετε ερωτήσεις ή σχόλια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να ευχαριστήσω και πάλι την Κομισιόν, διακόπτει ο Πρόεδρος και μπορούμε να πάμε στα διάφορα. Έχουμε τίποτα για τα διάφορα. Αν όχι, να ολοκληρώσουμε αυτή την ιστορική συνεδρίαση της Επιτροπής μας, λόγω ακριβώς της πληροφορίας για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα 5 λεπτά και θα συνεχίσουμε με τους συντονιστές σε 5 λεπτά. Μόλις γύρισε δηλαδή ο κύριος Δεκάστρο. Σε πέντε, πέντε λεπτά διάλειμμα. Ευχαριστώ.